Dear colleagues, we will start our today's meeting. Please sit down. Ας αρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Πολλά από τα μέλη της Επιτροπής μας είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε με την μεγάλη αντιπροσωπεία για τις Ηνωμένε Πολιτείε και ο κύριος δηλαδή ο πρόεδρός μας. Τον αντικαθιστώ λοιπόν σήμερα. Γι' αυτό ίσως και λείπουν εξέχοντα μέλη της Επιτροπής μας από τη σημερινή συνεδρίαση. Πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης χωρίς αλλαγές. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτον, για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα λάβει χώρα στις 26 Μαρτίου, το πρωί όμως μόνο. 26 Μαρτίου το πρωί, όχι το απόγευμα. Η απογευματινή συνεδρίαση ακυρώθηκε. Θα έχουμε και συνάντηση από κοινού με την Επιτροπή Άγκρη για τον φάκελο κλωνοποίηση. Στα πλαίσια του φακέλου αυτού λοιπόν που συνεργάζονται η Ένβη και η Άγκρη βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού η επόμενη κοινή τέτοια συνεδρίαση όπου θα συζητηθεί το σχέδιο έκθεσης για την κλωνοποίηση θα λάβει χώρα την 5η 16 Απριλίου 11 με 12 και 30. 16 Απριλίου λοιπόν, 11 με 12 και 30. Άλλη ανακοίνωση που έχω είναι ότι η διερμηνία στη σημερινή συνεδρίαση διατίθεται σε 22 γλώσσες. Δεν έχουμε εστονικά και γκέλικ. Ο ήθιστε υπάρχει μετάδοση στο διαδίκτυο βάσει της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Και περάμε στο τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμούσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε διαπραγματεύσεις για την τροπολογία όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων και την οδηγία σχετικά με την πρόθεση της χρήσης ενέργειας από ανανόσιμες πηγές στην πρώτη τρεμερή συνάντηση που έγινε τη 3η 10 Μαρτίου στο Στρασβούργο, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις για τις θέσεις τους. Επικεντρώθηκαν κυρίως στα βασικά πολιτικά ζητήματα. Πρόκειται για τους παράγοντες ήλου, χρήση ζής κτλ. Πρόκειται για τα αέρια του θερμοκηπίου, πρόκειται για το κάπινγκ, το όριο δηλαδή όσον αφορά την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων από ανανόσιμες πηγές ενέργειας και στόχους για ενέργεια, για ενέργεια από βιοκαύσιμα στις μεταφορές. Όλοι τόνισαν ότι πρέπει οι διαπραγματεύσεις να γίνουν με ανοιχτό πνεύμα, δεν εκπλήσει κανέναν αυτό. Και αυτό μάλιστα στα πλαίσια του γεγονότος ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο με την δεύτερη ανάγνωση. Ένας δεύτερος τριμερής διάλογος έχει προβλεφθεί για την 3η 24 Μαρτίου. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και παλήθευση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 525 κάθετος 2013. Η πρώτη ανάγνωση, θέση πρώτης ανάγνωση του Συμβουλίου συνάδει με τα σχόλια του συγητή που λέει να τη δεχτούμε τη θέση αυτή χωρίς παρετέρω τροπολογίες. Το χρονοδιάγραμμα είναι ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 26 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Απριλίου. Όσον αφορά τώρα την ε, μείωση της χρήσης σακουλών, πλαστικών σακουλών. Η ίδια κατάσταση. Η θέση πρώτης ανάγνωση του Συμβουλίου συνάδει με τις αποφάσεις της δικές μας, οπότε και εδώ η συγγήτρια προτείνει να το δεχτούμε χωρίς παρετέρω τροπολογίες. Το χρονοδιάγραμμα για το, για το θέμα αυτό είναι ότι ψηφίζουμε στις 31 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου πάλι. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις από αυτόν, τότε συνεχίζουμε και περνάμε στο σημείο 6. Πρόκειται για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μας ενημερώσει, να ενημερώσει την Επιτροπή μας για την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντζεγιάν Ρις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα την πρόταση αυτή κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η ιστορία της νομοθεσίας αυτής αρχίζει το 1965. 50 χρόνια δηλαδή ζωής έχει ο κανονισμός αυτός. Οι διατάξεις αυτές βέβαια συνδυάζονται και με άλλες πράξεις σχετικές στον κτηνιατρικό τομέα. <coughs> Ξέρουμε βέβαια ότι πολλές φορές ε, τα ακτινιατρικά φάρμακα ακολουθούν ε, αντίστοιχους κανόνες με τα φάρμακα για ανθρώπινη κατανάλωση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες αναφέρονται στον κανονισμό. Είναι και αυτό σημαντικό. Να το ξέρουμε. Ας δούμε λίγο το ιστορικό της νομοθεσίας αυτής. διαπιστώνουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Πότε αρχίσαμε δηλαδή. Αρχίσαμε λοιπόν το 2009 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε τον χάρτη πορείας. Στη συνέχεια είχαμε έκθεση των συμβαλωμένων, το 2011 ολοκληρώθηκε, είχαμε διαβούλευση, συναντήσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, το 2011, πιο στοχευμένες διαβουλεύσεις το 2012, το 2013 είχαμε πρώτη αξιολόγηση και το 2014 είχαμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της στις 10 Σεπτεμβρίου του 2014. Αν δούμε τώρα την νομική υφή της πρότασης αυτής. Πρόκειται για κανονισμό, αυτό προτείνουμε. για να μπορέσει να υπάρξει μια αναρμόνιση. Συμπεριλαμβάνουμε όλους τους κανόνες που έχουν να κάνουν με τα κτηνιατρικά προϊόντα σε έναν κανονισμό, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες υπάρχει ο κανονισμός 726 κάθετος 2004 για παράδειγμα. Θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια πιστεύουμε και θα υπάρξει και συμπλήρωση από κατεξουδιώτηση και εφαρμοστικές πράξεις. Προβλήματα. Ο ορισμός. Η έκθεση αντικτύπου διαπιστώνει ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά τις άδειες για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και ένα δεύτερο πολύ βασικό ζήτημα είναι το θέμα της ε, μικροβιολογικής αντίστασης. Αντίσταση στα μικρόβια. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα για είδη που δεν είναι πολύ πολυπληθή. Πρόβλημα υπάρχει και όσον αφορά τη θεραπεία μερικές φορές άλλων ειδών που είναι πολυπληθέστερα. και άλλα προβλήματα και για τις δύο περιπτώσεις. Η αρμόδια επιτροπή που έχει στοιχεία για τον πληθυσμό των διαφόρων ειδών μας έχει δώσει στοιχεία και σχετικά με την κατανάλωση. Πρόκειται για χείρους, ε, πουλερικά και άλλα τα οποία θεωρούνται ε, μεγάλα είδη και υπάρχουν και ορισμοί για μικρότερα είδη. Υπάρχουν επιπτώσεις εξαιτίας της έλλειψης φαρμάκων για τέτοια είδη, για τα λεγόμενα μικρά είδη. Αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες στην κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια. Το πλαίσιο οικονομικό που είχαμε μέχρι τώρα δεν απέτυχε σε όλα, χρειάζεται όμως σίγουρα ανακαίνιση. Χρειάζεται διόρθωση και συμπλήρωση. Επιτρέψτε μου να έρθω τώρα στους στόχους του κανονισμού αυτού. Να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών προϊόντων. Δεύτερον, να μειωθεί το διοικητικό άχθος. Τρίτον, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Τέταρτον, να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και τέλος, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους δημόσιας υγείας από την αντιμικροβιολογική αντίσταση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν και συγχρόνως διασφαλίζεται και η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η ασφάλεια τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να καλύπτονται από μια ενημερωμένη νομοθεσία Χρειάζεται αναθεώρηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Χρειάζονται περισσότερα κτηνιατρικά φάρμακα. αυτό είναι ο στόχος της αναθεώρησης. Δύο παραδείγματα σας αναφέρουμε εδώ. Το πρώτο έχει να κάνει με παντό είδου κτηνιατρικά φάρμακα, τα οποία θα μπορούν να έχουν ευρεία αδειοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει μια κεντρικής διαδικασία. κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Προτείνουμε επίση περισσότερα κίνητρα προς τη βιομηχανία για να αναπτύξει προϊόντα, κυρίως για τα μικρά είδη. Άλλες ε, διατάξεις προτείνουν περισσότερη ευελιξία για την χρήση των εκτινιατρικών ε, φαρμάκων εκτός συστήματος ε, αδειοδότησης. Προσπαθούμε επίσης να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Το επίπεδο προστασίας πρέπει να είναι ανάλογο με τα ωφέλη από την καινοτομία. Κίνητρα επίσης για επενδύσεις, ιδίως για μικρές αγορές, για μικρά είδη, για τις μέλησες όλους ιδιαίτερως. Αλλά όσο περισσότερο χρειάζεται να περιμένει κανείς ε, για να αποδώσει μια επένδυση, βέβαια τόσο πιο δύσκολο είναι να βρεθούν οι επενδυτές. Έχουμε καθορίσει 10 χρόνια ως στάνταρτ περίοδο, 14 χρόνια με δυνατότητα να υπάρξει επέκταση ένα χρόνο για τα μικρά είδη και επέκταση 4 χρόνια για τα μικρότερα είδη. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Έχουμε μέλισσες και χθείς με 13 χρόνια ανώτατη προστασία των προϊόντων και επέκταση η δεύτερη κατηγορία που για τα δόδημα ήδη. Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα μια ευκαιρία επίσης που λέει ότι μετά τα πέντε χρόνια αφού δοθεί η αρχική διαδότηση της αγοράς, ε, μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία. Εδώ βλέπετε τα περί καινοτομίας. Έχουμε έναν ότατο 18 χρόνια, ενώ για το μέλη της μέλισσας ή άλλα είδη υπάρχει συνδυασμός δυνατοτήτων. Η νέα πρόταση, η έτσι πρέπει να είναι τρία χρόνια πριν την ε, επέκταση. Έτσι οι επενδυτές μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα τη δουλειά τους. Προκειμένου τώρα να έχουμε ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, Προτείνουμε να διευκρινίσουμε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Σήμερα περιλαμβάνονται νέα είδη φαρμάκων, νέες θεραπείες για παράδειγμα, γιατί έχουν αναπτυχθεί τέτοιες τελευταία με, με τα βλαστοκύτταρα και άλλες περιπτώσεις και όσο περνά ο καιρός θα γίνουν περισσότερα θεραπείες ρουτίνας. Επίσης, οι νέοι ορισμοί βοηθούν όσον αφορά την αντιμικροβιολογική αντίσταση, τις δοκιμές ή τις περιορισμένες αγορές. Έπειτα έχουμε τις κλινικές δοκιμές. Θέλουμε να υπάρξει με τον κανονισμό αυτό μια μεγαλύτερη ομοιομορφία. Προτείνουμε επίσης την ε, τις διαδικασίες, οι διαδικασίες αυτές να γίνονται γνωστές βάσει μιας βάσης δεδομένων όπου όλα τα διαδοτημένα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλαμβάνονται. Άλλη στόχη του κανονισμού αυτού τώρα. Μείωση του διοικητικού άχθους. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε το διοικητικό ακριβώς άχθος. Για 538 εκατομμύρια το χρόνο για την φαρμακοβιομηχανία. 13% είναι ο τζίρος. Πολύ. Αλλού είναι 2%. Αυτό έχει να κάνει με τη σήμανση, με τις συσκευασίες. 184 εκατομμύρια βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Συζητήσει για νέες αγορές επίσης έχουμε μεγάλο κόστος. Προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άκθος λοιπόν για τις επιχειρήσεις και για τις αρμόδιες αρχές, η πρόταση συμπεριλαμβάνει διάφορες απλοποίησεις που δεν θα επηρεάσουν την ασφάλεια των κτηνιατρικών φαρμάκων. Πρώτον, οι άδειε στην αγορά άπαξ και χορηγηθούν δεν έχουν χρονικό όριο, ενώ σήμερα είναι μόνο για πέντε χρόνια. Δεύτερον, προτείνουμε απλοποίηση των κανόνων όσον αφορά τη συσκευασία και τη σήμανση. Δεν καθυστερούμε, ούτε αποκρύπτουμε καμία πληροφορία. Αλλά πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στα πακέτα. Και τρίτον, προτείνουμε και ένα νέο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης είναι κάτι που σήμερα θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογο στο τρέχον σύστημα. Αυτή η φαρμακοεπαγρύπνηση θα αντικατασταθεί, μέχρι τώρα υπήρχε για όλα, τώρα θα πηγαίνει αναφάκελο. Η πρόταση ακολουθεί την προσέγγιση κινδύνου ωφέλους. Και περιοδικά θα γίνονται ανανεώσεις των κανόνων αυτών. Θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα συνδυάζεται με την εισαγωγή κάποιων σημάτων που πιστεύουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό. Οι αρμόδιες αρχές με το σύστημα αυτό σε εθνικό επίπεδο θα ελέγχουν συλλογικά στοιχεία από κοινού και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προϊόντα. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα νέο, πιο αποτελεσματικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης που θα είναι πιο στάνταρτ και που θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μειώσουμε έτσι το άχθος κατά 47 δις το χρόνο. 2. Τώρα θα έρθω στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Βάσει των δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για την ε, σύνταξη της πρότασης, υπάρχει διαφορά στη δημιουργιανική των εκτινιατρικών φαρμάκων μεταξύ των ε, κρατών μελών. 30% της τιμής για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση καλύπτει και συμπεριλαμβάνει πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων διατάξεις για την έγκριση των, ε, ε, των πολιτών λιανικής στην εσωτερική αγορά. Αυτή δεν θα δίδεται σε ε, επίπεδο εθνικό. Θα δίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε μια ομάδα εγκεκριμένων πολιτών λιανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα εγκριθούν και οι πολιτές αλλά και οι πωλήσει θα επιτρέψουν την πρόσβαση στα κτηνιατρικά φάρμακα. Δεύτερον, προτείνουμε οι συνταγέ για τα κτηνιατρικά φάρμακα να αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ισχύει αυτό για τα φάρμακα για την κατανάλωση από ανθρώπου. Θα υπάρχουν ελάχιστε προδιαγραφέ για τι συνταγέ Έπειτα, Κατά τρίτον, ε, θέλουμε παρόμοια προϊόντα ε, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκριθούν με τον ίδιο τρόπο για την ίδια περίοδο ισχύω και απόσυρσης. Και να ολοκληρώσω με μια από τις πιο σημαντικές ε, διατάξει του κανονισμού, η μικροβιακή αντοχή και τα σχετικά μέτρα. Σήμερα, στις οδηγίες που ισχύουν, δεν υπάρχει διάκριση στην νομοθεσία μεταξύ των αντιμικροβιακών και άλλων ιατρικών φαρμάκων. Προτείνουμε συγκεκριμένε προδιαγραφέ για τα αντιμικροβιακά κτηνιατρικά φάρμακα, φάρμακα με ε, μια προσέγγιση που να βασίζεται σε επιστημονικέ γνώσεις. Έχουμε ένα κατάλογο διατάξεων εδώ προτινόμενων μέτρων για την, αντι, για την μικροβιακή ε, αντοχή. Θα αναφέρω μερικά. Υπάρχουν πολλά θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε κάποια αντιμικροβιακά μόνο για τους ανθρώπους, αλλά τα κάτι μέλη θα διασυνδέσουν τα δεδομένα τους για τα κύτταρα και τη χρήση των αντιμικροβιακών. Όλα τα αντιμικροβιακά φάρμακα θα πρέπει να συνταγογραφούνται εφόσον δεν ισχύει κάποιο ειδικό κανόνα. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να αρνηθούν την εμπορία των φαρμάκων ε, των κτηνιατρικών συγκεκριμένα εάν κάποιο αντιμικροβιακό είναι σε ειδική κατηγορία. Σας ευχαριστώ και θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρίς για αυτή τη διεξοδική περιγραφή της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των στόχων της και τώρα να ακούσουμε την εισηγητριά μας, την κυρία Γκροστέτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την άριστη παρουσίαση. Ιδιαίτερα λεπτομερή για την αναθεώρηση του κανονισμού, νομίζω η πρόταση της Επιτροπής συνολικά οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να μας επιτρέψει να ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει, δηλαδή τη διάθεση των κοινωνικών φαρμάκων. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με την διθεσιμότητά ε, τους μέσω της καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας από το τομέα την μείωση του διοικητικού άχθους και αυτό εντοπίστηκε σωστά, την βελτίωση των, ε, της αγορά αγοράς και την ε, καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Εδώ να σας αναφέρω και εγώ τα πρώτα μου σχόλια ε, τα πρώτα μου σχόλια του θέματος, να αρχίσω για την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιωτικά. Τα την μικροβιακή δηλαδή αντοχή. Ανέφερε 12 νέε διατάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σκοπό έχουν να ασχοληθούν με αυτό το μεγάλο ζήτημα. Νομίζω όμω ότι μπορούμε να πάμε πιο πέρα σε κάποια ορισμένα σημεία. Λόγω χάρη θα ήθελα να οριστεί η χρήση, η θεραπευτική, η μεταφυλακτική και η προφυλακτική των φαρμάκων και να απαγορευτεί η προφυλακτική χρήση των αντιβιωτικών. Δηλαδή χρήση μόνο για σκοπούς πρόληψης αυτό καλό θα ήταν να μην υπάρχει. Και το κείμενο ε, για τα προϊόντα, τα φαρμακευτικά, είναι κάτι που θα πρέπει να το αντικατοπτρίζει. Έπειτα στην έκθεσή μου διευκρινίζω και το εξή. Συνθήκε εντό των οποίων οι επαγγελματίε του τομέα τη υγεία, την ίαντρη δηλαδή, έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν και να πολλούν αντιβιωτικά. Ξέρουμε ότι εδώ κάποιε πρακτικέ ε, μεταξύ των κρατών μελών διαφέρουν τρομερά. Ε, Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια πρόταση που να μπορεί να γίνει αποδεκτή και να μπορεί να είναι και εφαρμόσιμη από το σύνολο των κάτω μελών. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω για αποσύνδεση όπως θα το ήθελαν κάποιοι, ε, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ε, τεράστιες πρακτικές δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε στο άρθρο 107 την έννοια ζώα που μπορεί να ε, περιθάρει ο κτηνίατρος αγωγή προς ζώα, αυτό εντό εισαγωγικών πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μετά την διάγνωση, την ε, κλινική δοκιμή και την διάγνωση, οπότε εφόσον ε, διαπιστωθεί ότι ένα ζώο ε, είναι ασθενή, εκεί θα πρέπει να διευκρινίζεται αυτό πολύ ξεκάθαρα. Η Επιτροπή επίσης θέλει ένα κατάλογο αντιβιωτικών, κρίσιμων αντιβιωτικών, που θα προορίζονται μόνο για την ανθρώπινη χρήση. Αυτό το βρίσκω ενδιαφέρον. Το στηρίζω. Αυτή τη στιγμή όμω ο κατάλογο αυτό βασίζεται σε κριτήρια αυστηρό επιστημονικά. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχει συντάξει συγκεκριμένε συστάσει επί του θέματο. Μου φαίνονται πολύ εύστοχε και καλό να τι ακολουθήσουμε. Τέλο. Και εδώ θα διαφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι η επιγραμμική πώληση αντιβιωτικών είναι αρκετά επικίνδυνο. Ναι, εντάξει, δεν λέω, πρακτικό ακούγεται. Αλλά δεν υπάρχει πλέον κανένα έλεγχο για τη χρήση των αντιβιωτικών αυτών. Για την ποιότητά του επίση. Οπότε νομίζω ότι η πώληση στο διαδίκτυο όχι μόνο των αντιβιωτικών αλλά και των συνταγορφημένων κτηνιωτικών φαρμάκων, ε, ε, έχει σοβαρότατο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό θα έλεγα καλό να είναι να απαγορευτεί αυτό. Εδώ θα διαφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και θα είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ελπίζω να έχω τη στήριξη και των υπολοιπών συναδέλφων για το θέμα αυτό. Τώρα, το θέμα της καινοτομίας και της έρευνα Η αγορά των δυνατικών φαρμάκων είναι όντως σχετικά μικρή. Είναι κατακαιρματισμένη φαρμακοβιομηχανίε δεν έχουν ενταρρυνθεί να προχωρήσουν στην κοινοτομία και να ε, θέσουν σε πορεία νέα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν η καινοτομία να υποκινηθεί, γι' αυτό χρειάζονται και μέτρα ενθάρρυνσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιο βαθμό το κάνει αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό να είμαστε λίγο φιλοδοξότεροι. Δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε μια όθηση στην καινοτομία στον τομέα αυτό, καλό θα ήταν και προτείνω η περίοδος ε, φύλαξης των δεδομένων όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο αυτή δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες αλλά 18 χρόνια μέγιστης προστασίας για τα νέα ε, αντιβιωτικά αντί για 14 ίσως να είναι μια λύση το να προβλέψουμε μια διετία επιπλέον προστασίας για κάθε πολιτικές είδος που καλύπτεται από αυτή την κατηγορία με έναν επιπλέον χρόνο παράτασης και αυτό ίσως να είναι μια λύση, αλλά θέλω να επανέλθω στην απαγόρευση των ζώων ε, με κλινικέ δοκιμέ που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένε προθεσμίες που τηρούνται και ισχύουν. Δεν υπάρχει λόγο για αυτή τη διάταξη, δεν έχει λόγο ύπαρξη η διάταξη αυτή. Αρκεί να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό αυτών των διατάξεων. Η Επιτροπή αναγνώρισε και ίσω να πρέπει αυτό να το συζητήσουμε μέσω τη έκθεση. Αναγνώριζα ότι εδώ μπορεί να μην είναι ακριβώ έτσι. Για την φαρμακοεπαγρύπνηση έκανε μια άριστη πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να περιοριστεί το διοικητικό άχθο. Είναι σημαντικό. Η σημερινή διαδικασία είναι όντω ε, περίπλοκη και θα πρέπει ε, τέλει να επιμείνουμε σε ένα σύστημα φαρμακοεπαγρύπνηση που να βασίζεται στην, ε, στον εντοπισμό του κινδύνου. Αυτή την προσέγγιση την επιθυμώ και εγώ, αλλά δεν θα ήθελα να πλήξουμε την δημοσία υγεία σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τη σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη ασφάλεια που προσφέρει η φαρμακοπαρύπνηση και την ε, προστασία της δημόσιας υγείας. Πρέπει αυτή η ισορροπία να βρεθεί και να βασιστούμε και στην ε, συστηματική ε, αξιολόγηση του κινδύνου και της ωφελίας που προσφέρει ένα προϊόν στα πρώτα χρόνια της ζωής του τουλάχιστον και μετά κίνδυνο και την ε, ανείχνευση ε, ενδεχομένων επιπτώσεων. Η Επιτροπή το ανέφερε στην παρουσίασή της, το ανέφερε και μας φώτισε και αυτό το νέο σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης, αλλά καλό θα να διευκρινίσουμε κάπως. Όσο για τις διαδικασίες αδειοδότησης και θέσεις σε εμπορία, θέση στην αγορά, είναι σημαντικό να έχουμε μια ενιαία ε, έγκριση σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό είναι νομίζω το μέλλον. Θα πρέπει βεβαίως να κάνουμε μια προσπάθεια να οδηγηθούν προς τα εκεί οι μας, αλλά η αγορά των κτηνιατικών φαρμάκων δεν είναι η αγορά των ε, φαρμάκων για ανθρώπινη κατανάλωση. Υπάρχουν ακόμη πολλές ε, διαφορές και είναι αποκεντρωμένες ακόμη διαδικασίες που εφαρμόζονται. Και εδώ Καλό θα ήταν να βρούμε μια θέση που ίσως να μην είναι ιδανική, αλλά θα μπορούσε να στηριχθεί από τους περισσότερους. Κάποιες βελτιώσεις ίσως λοιπόν να μπορούν να επιφερθούν για να βελτιώσουμε και άλλο, και άλλο αυτές τις διαδικασίες και την πρόσβαση σε αυτές. Όσο για την προστασία του περιβάλλοντος, σίγουρα οι μελέτες αντικτύπου για το περιβάλλον είναι πολύ χρήσιμες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια σειρά από για την επικαιροποίηση όποτε αυτό χρειάζεται. Καλό θα ήταν να πάμε και λίγο πιο μακριά. Αλλά το όλο σύστημα είναι ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικές οι μονογραφίες, δηλαδή μελέτες αντικτύπου, όχι αναπροϊόν, αλλά αναμοριακή σύνθεση. Έτσι θα προστατεύονται τα δεδομένα που περιλαμβάνουν αυτέ οι μελέτε που είναι και ιδιαίτερα δαπανηρέ για τι φαρμακοβιομηχανίε, αλλά τουλάχιστον έτσι θα υποχρεωθούν οι φαρμακοβιομηχανίε να ενώσουν τι δυνάμει του, να λειτουργήσουν ω ομάδα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι οδεύουμε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα περιορίσει και το, το σημαντικό κόστο. Ξέρω βεβαίω ότι αυτέ οι μονογραφίε είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Το σκέφτομαι το όλο θέμα και θα ήθελα τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματο. Υπάρχουν πολλέ άλλε λεπτομέρειε που θα μπορούσα να θίξω, γιατί η πρόταση και η παρουσίαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ήταν διεξοδική, όμω δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είναι σημαντικό να ακούσουμε και του πιο συζητητέ και να δούμε πώ θα τοποθετηθούν για τα σημαντικότερα αυτά ζητήματα με τα χαράς να ακούσω τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσουν τώρα οι σκιώδεις συζητητές. Δεν θέλω να σας ε, αγχώσω. Έχουμε χρόνο. Αλλά παρακαλώ τους ε, σκιώδεις παρόλα αυτά να είναι συνοπτικοί. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ή δυνατόν. Πρώτον, ο σκιώδης των σοσιαλιστών, ο κύριος Τανασέσκου. η πρόταση για αυτά τα νέα μέτρα, τα νομοθετικά, είναι ένα βήμα προς την ε, ενιαία αγορά. Διότι επεκτείνεται η συγκεντρωτική διαδικασία αδειοδότησης, μία βάση δεδομένων που θα περιέχει όλα τα εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα, την εναρμόνιση των συνοψίσεων των ε, χαρακτηριστικών, τα υγειονομικά και φυτογειονομικά και άλλα. Αν ε, έχουμε όμως ε, μια παράταση και των άλλων δυνατοτήτων αδειοδότησης, μπορεί να είναι μια λύση για τις φαρμακοβιομηχανίες που δεν έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για αυτή τη συγκεντρωτική ε, αδειοδότηση ή για προϊόντα περιορισμένης αγοράς. Βεβαίως και η πρόταση για την έγκριση των κλινικών δοκιμών, για την αρμόνιση που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει είναι θετική, η προθεσμία είναι 60 ημέρες για την έγκριση των δοκιμών. Αυτό ήταν απόλυτα αναγκαίο, ούτω ώστε τα προγράμματα ανάπτυξης νέων φαρμάκων δεν καθυστερούν περιμένοντας την έγκριση των δοκιμών. Αυτό που με ανησυχεί ωστόσο <clears throat> είναι η επίπτωση στην πράξη της αφαίρεσης ε, της δυνατότητας να αποσύρονται ορισμένα προϊόντα στα πλαίσια των δοκιμών. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ζώα που θα συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές και στα οποία θα δίδονται αυτά τα νέα προϊόντα, δεν μπορούν να μπουν στην ε, διατροφική αλυσίδα, ακόμη και αν μπορέσουμε να αποτιμήσουμε ότι ο κίνδυνος για τον καταναλωτή είναι αποδεκτός. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα πολύ ισχυρό αντικίνητρο για την ανάπτυξη νέων κτηνιατρικών φαρμάκων και ενδεχομένω λοιπόν και νέων κατηγοριών αντιμικροβιακών. Χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν για την συσκευασία και τη σήμανση ότι πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν αυτές οι απλωστευμένες πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτω ώστε να υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση για τους χρήστες και βεβαίως να είναι σαφή και επανάγνωστα αυτά τα στοιχεία. Αν είναι υπερβολικά υπερβολικές οι απαιτήσει ε, για πληροφόρηση τότε ε, είναι όντως αυτό σοβαρό, σοβαρή τροχοπέδιο, όπως έχω αναγνωρίσει για την ε, εισαγωγή νέων φαρμάκων. Πρέπει όμως να επιτρέψουμε στις εταιρείες αν θέλουν να προσθέσουν ε, πληροφόρηση για λόγους ασφαλείας στη συσκευασία χωρίς ωστόσο αυτό να είναι υποχρεωτικό. Αυτή η συμπροματική πληροφόρηση πρέπει να αναλύεται από το φορέα ή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όταν υποβάλλεται αίτηση για ε, εμπορία των φαρμάκων αυτών. Για τη σήμανση, για το, τη δυνατότητα ε, επιστροφής μπορεί να έχει πρόβλημα λόγω των διαφορετικών διατάξεων στα κράτη-μέλη. Για λόγους ασφάλειας και για περιβαλλοντικούς λόγους πιστεύω ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί αυτό το σύστημα επιστροφής. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι τμήμα της πρότασης αυτής που κάνουμε τώρα για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η πρόταση αυτή επίσης δεν ασχολείται με τις προτεραιότητες που υπάρχουν για να προστατεύουμε επαρκώς το περιβάλλον από τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τι χρειαζόμαστε όχι να κάνουμε νέα αποτίμηση πολλών προϊόντων, αλλά να έχουμε επαρκή στοιχεία για τις επιπτώσεις των περιβάλλων, των ενεργών ουσιών των κτηνιατρικών φαρμάκων που ξέρουμε ότι αποτελούν, αποτελούν κίνδυνο. Έχουμε ήδη παραδείγματα σε άλλα ενωσιακά νομοθετήματα για την ε, ε, διάδοση πληροφόρησης μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και σε αυτό το μέτρο αυτό θα προωθούσε και την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία. Επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε σε αυτή την πρόταση πώς θα γίνεται ο έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα γενώσιμα. Για να μην έχουμε επικάλυψη και μελέτες που δεν προσφέρουν τίποτα όσον αφορά την πραγματική μείωση του κινδύνου. Είμαι υπέρ της εναρμόνισης των υγειονομικών και φυτο-υγειονομικών SPS αλλά αυτό που προτείνεται δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα εναλλακτικό σύστημα. Αυτά που περιέχει τώρα η πρόταση για ε, τη χρήση πέρα από τους όρους της πρότασης αυτής, για λόγους για παράδειγμα αντιμικροβιακής ε, αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής θα πρέπει να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουμε ε, όταν υπάρξουν νέα αντιβιωτικά. Γιατί αυτό θα επηρεάσει και τους ε, κτηνιάτρους το τι αντιβιωτικά να προτείνουν. Έχω επιφυλάξει και για το παλιό σύστημα, το σύστημα χιονοστιβάδα. Γι' αυτό θα προτιμούσα ένα μεικτό σύστημα. Για το θέμα των ε, πωλήσεων στο ίντερνετ για κτηνιατρικά φάρμακα. Βεβαίως, πολύ καλή αυτή η πρόταση, αλλά φοβάμαι ότι η πρόταση αυτή δεν περιέχει επαρκείς διατάξεις για να ελέγχουμε επαρκώ το περιβάλλον. Ιδιαίτερα για τις πωλήσει αντιμικροβιακών. Η συλλογή στοιχείων για το τι πωλήσει γίνονται και για τη χρήση αυτών των αντιμικροβιακών κτηνιατρικών μπορεί να μην είναι όπως έχει τώρα η πρόταση. Συνολικά, η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών σε όλη την Ένωση. Και λόγω των ιδιομορφιών της αγοράς αυτής πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την προστασία τεχνικών στοιχείων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, για νέα είδη ή για νέες χρήσεις. Καλωσορίζω τις βελτιώσεις για το σύστημα φάρμακοεπαγρύπνησης, γιατί έχουμε καλύτερη χρήση των πόρων και αντιμετώπιση και των κινδύνων που προκύπτουν από αυτά τα προϊόντα και αυτό τον κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τανασέσκου. Ο, ο κύριος Μπίχα που είναι σκιώδης του ε, ECR. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική αυτή η προσπάθεια για να έχουμε ένα νομοθέτημα για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Είναι αρχικό κείμενο αυτό, άρα χρειαζόμαστε μερικές ε, εξηγήσεις, όχι μόνο τροποποιήσεις. Το πρώτο είναι τι επίπεδο ασφάλειας έχουμε. Γιατί το κείμενο αυτό λέει ότι θέλει να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας και των ζώων και των ε, ανθρώπων. Κάποιες διατάξεις ιδιαίτερα αυτές που μειώνουν τις προϋποθέσεις για τις εταιρείε. Μειώνονται κατά πολύ λοιπόν οι υποχρεώσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και επίσης ε, αποδυναμώνονται και κάποιες ε, διατάξεις για την εμπορία. Άρα πώς αυξάνεται, δεν νομίζω ότι αυξάνεται η ασφάλεια. Αντίθετα νομίζω ότι μειώνεται. Κάτι άλλο που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Η Επιτροπή βλέπω ότι γράφει ότι τα κτηνιατρικά είναι σχετικά ακριβά. Οπότε η Επιτροπή λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι τιμές με βάση τον νέο αυτοκανονισμό. Αλλά αυτά που βλέπουμε εδώ να αναφέρεται για την καινοτομία. Η καινοτομία πάντα δημιουργεί προβλήματα, είναι επίμαχη, αλλά είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα για να έχουμε νέα αντιβιωτικά. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ καιρό τώρα επαναλαμβάνει το ίδιο τροπάριο ότι οι περίοδοι προστασίας των δεδομένων είναι πολύ εκτεταμένες άρα πρέπει να μειωθούν. Να έχετε υπόψη σας ότι οι τιμές ε, των φαρμάκων συνδέονται κατά πολύ με το πόσο γρήγορα ε, μπαίνουν στην αγορά τα γενώσιμα. Τα μέτρα λοιπόν που προτείνεται δεν νομίζω ότι θα μειώσουν τις τιμές. Μπορούμε έτσι να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Όχι. Με άλλο τρόπο. Σκεφτόμαστε μόνο τη δημιουργία προτύπων και τις ε, διατάξεις ε, για τα, την ευρεσιτεχνία. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Διαβάζοντας αυτό το σχέδιο μου δημιουργείται η εντύπωση ότι η διανομή των κτηνιατρικών φαρμάκων ιδιαίτερα ε, αυτών που όντως θα χρησιμοποιήσουν ε, οι ε, γεωργοί επί των ζώων λέγεται ότι θα τα χρησιμοποιήσουν επίσης οι ειδικοί για τα ζώα. Τι πάνε για τα ζώα. Δεν είναι κτηνίατροι είναι αυτή η νέα ορολογία. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη. Θα θέλαμε για παράδειγμα για την χρήση ε, φαρμάκων στους ασθενείς να λέμε ότι θα τα χρησιμοποιούν και θα τα συνταγογραφούν κάποιοι ειδικοί για την υγεία αλλά όχι γιατροί. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Ανοίγουμε παράθυρα ούτω ώστε ε, να υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί που δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Στο σχέδιο κανονισμού τίθενται πολλά θέματα, πολλά θα συζητηθούν. Θα υποβληθούν πολλές τροπολογίες, θα γίνουν πολλές διορθώσεις. Να αναφέρω μερικές λοιπόν και εγώ από τις επιφυλάξεις μου για αυτό το κείμενο. Μετά από μια πρώτη γρήγορη ανάγνωση στο άρθρο 104 υπό παράγραφος 3 Βλέπουμε να αναφέρεται ο όρος μικρές ποσότητες ε, κτηνιατρικό φαρμάκο. Τι είναι μικρή ποσότητα, 5 τόνι ή ένα γραμμάριο. Και αναφέρεται επίσης ο όρος ότι πρέπει να υπάρχει μια τριετής περίοδος διατήρησης κάποια τεκμηρίωσης, η οποία είναι όμως πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σε περιπτώσεις παρενεργειών ή άλλων ανησυχητικών επιπτώσεων ε, επί των ανθρώπων. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αλλων ανησυχητικων επιπτωσεων είναι επαρκής. Κάτι άλλο που με ανησυχεί. Πωλήσει ε, μέσω διαδικτύου. Βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντικό το ίντερνετ. Αλλά εάν μπορεί κανείς να αγοράσει στο ίντερνετ ε, την ιατρικά φάρμακα, ωραία. Αλλά τι έλεγχος υπάρχει. Πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε πού πάνε αυτά τα φάρμακα. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ουσιαστικός, αποτελεσματικός έλεγχος ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια και των ζώων και των ανθρώπων. Που είναι θέμα κλειδί για το όλο θέμα. Κάτι άλλο που πρέπει να μας εξηγηθεί καλύτερα είναι πώς γίνονται οι συνταγογραφήσεις. Τι πρέπει να περιέχουν οι συνταγές. Τι βλέπουμε εδώ να λέει. Λιγότερη γραφειοκρατία. Άρα λιγότερη πληροφόρηση. Και θα είναι όπως ξέρετε πανευρωπαϊκή η αδειοδότηση. Θα έχουμε κάποια στάνταρ ε, κάποια στάνταρ πληροφόρηση που θα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτά προκατακτικά μόνο από πλευρά μου. Νομίζω ότι πολλά μπορούμε να πούμε ακόμη και καταλήγοντας Θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε όλες αυτές τις σημαντικές πλευρές του θέματος αυτού σε ένα μόνο κείμενο, γιατί ξέρουμε ότι Η μη ορθή χρήση ε, των ε, κτηνιατρικών μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συντονισμένη ε, αντιμετώπιση και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ για λόγους ευγένειας και προς τους άλλους συναδέλφους να τηρείτε το χρόνο σας. Πέντε λεπτά. Σκιώδης Άλντε. Η κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτέλους ήρθε και μας παρουσίασε την πρόταση αυτή. Πράγματι, βλέπετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Επιτροπές του Περιβάλλοντος και Γεωργίας ήδη από το 2011 και το 2012 είχε απαιτήσει να συνταχθεί, να εκπονηθεί ένα τέτοιο έγγραφο, κυρίως για τα αντιβιωτικά που δίνουμε στα ζώα. Το 90% είναι προτάσεις της κυρίας Γκροστέτ. Στην πρόταση αυτή πιστεύω ότι οι ορισμοί δεν είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι λέμε σε όλους τους τομείς, σε όλα τα σημεία. Πρέπει να γίνει απλοποίηση λέμε, ναι βεβαίως, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχουν τέσσερις τρόποι, πολύ περίπλοκοι, για να πάρει άδεια ένα νέο κτηνιατρικό φάρμακο. Αφού λέμε ότι θέλουμε να απλοποιήσουμε. Οι υγειονομικές αρχές θα συνεδριάζουν, οι γιατροί θα συνεδριάζουν, θα υπάρχει μια ομάδα συντονισμού. Γιατί, γιατί να υπάρχει τέτοια επικάλυψη τέτοια γραφειοκρατία. Δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια διαδικασία κεντρική έγκρισης και σε εθνικό επίπεδο να είναι συμπληρωματικό το τι γίνεται για τις μικρές επιχειρήσεις ή για τις νέες, για τις startup οι οποίες ε, θα μπορούν να τυχαίνουν χειρισμού πιο κοντά θα έλεγα στις αρχές. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την ε, γραφειοκρατία. Χρειαζόμαστε περισσότερη απλοποίηση. Έπειτα ένα από τα ζητήματα κλειδί σήμερα είναι για την υγεία του κοινού, έτσι. Είναι η αντίσταση ακριβώς ε, στα αντιβιωτικά. Πολύ συχνά τα... τους όρους τους χρησιμοποιούμε εσφαλμένα, γιατί μιλάμε για αντίσταση στα μικρόβια, βακτηρίδια, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Η κυρία, η κυρία Γκροστέτ πάντως έχει δίκιο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά πριν να έχουμε τη διάγνωση. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τη χρήση αντιβιωτικών έτσι προληπτικά. Όχι. Άπαξ και έχουμε τη διάγνωση, τότε ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη διάγνωση από ένα κτηνίατρο και τότε μόνο να προσφεύγουμε στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δούμε πιο περιορισμένα αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά την συνταγογράφηση online, μέσω διαδικτύου δηλαδή, ανοσπιτικών φαρμάκων ή αντιβιωτικών, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και υπάρχει και κάτι που δεν καταλαβαίνω. Και ισχύει για πολλές χώρες αυτό. Έχουμε ειδικά φάρμακα, ειδικότητες γιατρών όταν πρόκειται για την ανθρώπινη υγεία. Οι άνθρωποι αυτοί φυσικά γνωρίζουν πολύ καλά τον κλάδο τους, τη δουλειά τους. Στην κτηνιατρική όμως, αυτό που ονομάζουμε κτηνίατρος, πανεπιστημιακά, έχει σπουδές αντίστοιχες με εκείνες των γιατρών για τους ανθρώπους, αλλά κάπου τον χρησιμοποιούμε απλώς για τη συνταγογράφηση. Δεν το θέλουμε πραγματικά γιατρό. Ενώ είμαι σίγουρη ότι ένας κτηνίατρος είναι ένας πραγματικός γιατρός. Δεν πουλάει μόνο κτηνιατρικά φάρμακα. Μπορεί να μου πείτε ότι είναι λεπτομέρεια, αλλά για μένα είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να συζητήσουμε και που πρέπει να τη βάλουμε και μέσα στο κείμενο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πόλσον και ευχαριστούμε που τηρήσατε το χρόνο σας. Γκουε τώρα. Η κυρία Κίλεν είναι σκιώδης. η συγκήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Ποιο είναι το σημείο κίνησης. Πρέπει να είναι πάντα η πρόληψη. Πριν χρησιμοποιήσουμε κτηνιατρικά φάρμακα. Ε, δυστυχώς όμως δεν είναι αυτό πάντα εφικτό. Υπάρχει και το θέμα της αντίστασης στα μικρόβια. Ένα ζήτημα που γίνεται όλο και πιο σημαντικό όσο περνά ο καιρός. Εδώ έχουμε διατάξεις για την ανάπτυξη κτηνιατρικών φαρμάκων και τη χρήση τους. Χρειαζόμαστε, πιστεύω, σαφείς διατάξεις όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων αυτών. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε μόνο διατάξεις για τη διάθεση στην αγορά, για την ανάπτυξη για τη διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊόντων. Όταν μιλάμε λοιπόν για την χρήση προϊόντων off-label, δηλαδή άρθρα 115 με 117, είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε τα γενώσιμα αυτά προϊόντα, τα off-label, με έναν κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος δηλαδή πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση αυτή των προϊόντων. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δούμε ποιες είναι οι αναλλακτικές λύσεις που έχουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χρήση των προϊόντων αυτών είναι ασφαλής για τα ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη της. Θα ήθελα όμως επίσης να ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σημείο. Τώρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ασφαλή χρήση των προϊόντων αυτών off-label, μιλάμε για ένα σύστημα χιονοστιβάδας. Εγώ νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε να έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία, ενώ στόχος των διατάξεων αυτών είναι η μείωση ακριβώς της γραφειοκρατίας. Τι γίνεται και με την παρακολούθηση της πώληση των οκτηνιατρικών προϊόντων. Είναι πάντα ένας κτηνίατρος που πρέπει να παρακολουθεί την πώλησή τους, κυρίως όταν αυτή γίνεται μέσω διαδικτύου. Αυτό θα είναι ευθύνη των χωρών μελών. Πάντως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι αναγκαία τα προϊόντα αυτά και ακολουθούν μια συνταγογράφηση. Ο κτηνίατρος μπορεί να πουλήσει κτηνιατρικά προϊόντα στους ε, κτηνοτρόφους. Αυτό είναι θετικό. Αλλά τα προϊόντα αυτά πρέπει να πολλούνται μόνο για τα ζώα που είναι στην αρμοδιότητα, είναι στην ευθύνη ακριβώς του συγκεκριμένου κτηνιάτρου. η χρήση του προϊόντος δηλαδή να είναι για συγκεκριμένα ζώα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την γραφειοκρατία είναι και το εξή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα και για τα οποία χρειάζεται άδεια, αλλά Θέλω να μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη. Τέλος, υπάρχει και το θέμα της εισαγωγής κτηνιατρικών προϊόντων και ταξινόμησή τους. Προτείνουμε κάτι που θυμίζει αυτό που έχουμε για τα φάρμακα. Δεν κινδυνεύουμε όμως να καταλήξουμε σε κακή χρήση των κτηνιατρικών αυτών προϊόντων. Ίσως πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το άρθρο. Πρέπει να αποφύγουμε τα κτηνιατρικά αυτά προϊόντα να καταλήξουν στον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χόσλινγκ, εκ μέρους των Πρασίνων και ορίστων των Πρασίνων. Αγαπητοί συνάδελφοι, με απογοήτευσε κάπως η πρόταση της Επιτροπής γιατί είχαμε τη δυνατότητα πιστεύω να αντιμετωπίσουμε το βασικό πρόβλημα που είναι η τρομερή κατάχρηση αντιβιωτικών στα κτηνιατρικά. Αλλά μόνο τελευταία στιγμή ασχολείται με αυτό το θέμα. Η Κομισιόν λέει περισσότερη ανταγωνιστικότητα, λιγότερη γραφειοκρατία, καινοτομία. Ναι, όλα αυτά καλά. Αλλά το βασικό είναι να μειώσουμε τη χρήση αντιβιωτικών. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν λέει τίποτα γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν. Πρέπει κάτι να επαναλάβουμε. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Κομισιόν, έχουμε 25.000 θανάτους το χρόνο λόγω αντίστασης στα αντιβιωτικά και έχει να κάνει και με τη χρήση αντιβιωτικών στα ζώα. 600 600 τόνοι, λέει ο μιλητή, χρησιμοποιούνται, αντιβιωτικών χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη χρήση και 1300 τόνοι για κτηνιατρική χρήση. Επίσης, κάτι άλλο που δεν ε, αναφέρεται στην πρόταση. Τι θα γίνει με τις επιπτώσεις των αντιβιωτικών μετά τη χρήση τους, για παράδειγμα, κατά την ε, πάχυνση των ζώων η χρήση αυτή υποτίθεται ότι απαγορεύεται, αλλά υπάρχουν τρομερές μη επιτρεπόμενες χρήσεις και ούτε προφυλακτικά είναι σωστή η χρήση τους, ούτε μεταφυλακτικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αν αρρωστήσει ένα ζώο σε ένα υπόστεγο, τότε δίνουμε σε όλα τα ζώα στο υπόστεγο αντιβιωτικά. Επίσης, ο ρόλος των κτηνιάτρων πρέπει να αντιμετωπιστεί κριτικά για ορισμένα σημεία. Διότι όπως υπόθηκε πολλές φορές ε, το εισόδημά τους το βγάζουν από την πώληση φαρμάκων οπότε έχουν συμφέρον να τα πολλούν για να κερδίζουν περισσότερα. Πρέπει και εδώ να δούμε τι περιορισμούς μπορούμε να εισαγάγουμε. Και επίσης με απογοητεύει ότι δεν αντιμετωπίσαμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των αντιβιωτικών και γενικότερα των κτηνιατρικών φαρμάκων. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε αντιβιωτικά και στο υπόγειο, στα υπόγεια ύδατα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο σημαντικό τμήμα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Και όπως είπαν όλοι σαφώς, Μέχρι τώρα, πωλήσει στο ίντερνετ δεν είναι δυνατόν. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την υπερβολική χρήση, πώς θα ελέγξουμε. Είναι τέλος λάθος. Και επίσης αυτή η απεριόριστη χρήση χρονικά, ε, συγγνώμη, η απεριόριστη αδειοδότηση χρονικά των ε, αντιβιωτικών για τα κτηνιατρικά. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν ε, ε, προθεσμίες και περίοδοι, γιατί εντωμεταξύ προκύπτουν νέες ε, επιστημονικές ανακαλύψεις. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Υπάρχουν ορισμένα τα λεγόμενα αντιβιωτικά τελευταίας, ως τελευταία, τελευταίας προσφυγής. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ιατρική. Αυτό είναι η τελευταία μας γραμμή αμήνης για τους ανθρώπους που έχουν αναπτύξει αντίσταση στα άλλα αντιβιωτικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ζώα. Πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμη. Πρέπει να θέσουμε θεμελιώδη ερωτήματα για, την, ε, για τους στόχους που έχει αυτό το νομοθέτημα. Πρέπει να υπάρξει ισχυρότερος έλεγχος για τη χρήση των αντιβιωτικών και να περιορίσουμε των ε, κτηνιατρικών και να περιορίσουμε τα αντιβιωτικά και μια τέτοια πρόταση δεν υπάρχει σε αυτό το κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Πεντιτσίνη από την ΕΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία πρώτη εντύπωση μετά από το σχέδιο αυτό κειμένου Φαίνεται σαν να ανοίγεται μπροστά μας ένα τεράστιο, ένας τεράστιος χώρος, σαν ένα λιβάδι που δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα αρκετά. Ένα ανεξερεύνητο πεδίο και δεν έχουμε ακόμη κάνει αρκετά για να αποκτήσουμε σχετικά γνώσεις. Στόχος των εταιριών είναι βεβαίως να υπάρχει ενιαία αγορά για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Ο δικός μας όμως θα πρέπει να είναι να διαφυλάξουμε την ευζοία των ζώων και βεβαίως την καλή υγεία των ανθρώπων. Και θα πρέπει να σκεφτούμε και την ε, περίθαλ, αγωγή ε, μαζικά, αλλά και για το καθένα ζώο ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν όπως έχει προγίνει η πρόταση μας δημιουργεί πολλούς ενδιασμούς. Μας φαίνεται σε σχέση με τις φαρμακοβιομηχανίες ε, να έχει σοβαρή έλλειψη ισορροπίας. Αρχίζει η δημιουργία μιας τεράστιας αγοράς με πολύ λίγους περιορισμούς και υπάρχουν κίνδυνοι και για την υγεία, για την ανθρώπινη υγεία. Συμφωνώ με τους σκιώδης εισηγητές, το, με τους των Τρασίνων, όταν λέει ότι ορισμένα υποθέσεις της πρότασης είναι τελείως αμφισβητούμενες. Δηλαδή, όντως είναι καλή ιδέα να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Πού είναι τα δεδομένα που δείχνουν ότι είναι θετικό να υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Από την άποψη της αγοράς εξυπηρετεί ή από την άποψη της ε, υγείας των ζώων ή των ανθρώπων. Και ισχύει αυτό για ολόκληρο τον τομέα ή ισχύει γενικώ, διότι πρέπει να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε ακριβώ. Έχουμε πολλού επιφυλάξει για την προφυλακτική χρήση των φαρμάκων και εδώ θα συμφωνήσω με του συζητητέ του Κοινοβουλίου και με τη συνάδελφο Πάουνσελ, διότι σε ποιε περιπτώσει θα πρέπει να κρίνεται η προφυλακτική χρήση και με, με ποιου κανόνε. Εδώ ε, περνάμε σε μια κατάσταση γεμάτη κινδύνου και για την ανθρώπινη υγεία. Είμαστε βέβαιοι ότι η απεριόριστη χρήση των αδειών ε, τη εξουσιοδότηση είναι καλή ιδέα. Μήπω ε, μετά περάσουμε σε μια μετάκλητη αλλαγή στην αγορά, εάν κάνουμε διαφορετικέ διαπιστώσει σε κάποια χρόνια στο μέλλον. Και με το off-label, πώ θα επιτραπεί αυτή η χρήση. Δεν μιλώ εδώ για γενώσιμα ή παρόμοια φάρμακα. Μιλάω για το off-label που υπάρχει συνταγή, αλλά το φάρμακο ξεπερνά τα όρια της συνταγής. Για κάθε φάρμακο υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη συνταγογράφηση βάσει του evidence-based management, αλλά το off-label ξεπερνάει την κλασική συνταγογράφηση. Αυτό είναι το off-label. Υπάρχει μετά και το θέμα της ομοιότητας ή της, του γενικού χαρακτήρα του φαρμάκου. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις και αν μιλήσουμε για γενώσιμα και παρόμοια φάρμακα, η ελεύθερη πώληση χωρίς δυσκολίες ε, των φαρμάκων αυτών ε, πώς θα οριστεί. Δεν είναι ότι είμαι αντίθετο, αλλά καταλάβαινα ότι η συγκέντρια του Κοινοβουλίου ήθελε να δώσει την εξής κατεύθυνση. Να εισάγουμε μία αδειοδότηση για το μόριο, τη μοριακή σύνθεση και όχι για το προϊόν ή την ε, εταιρεία, την μάρκα ε, και για τα πορίσματα της η πραγματική καινοτομία θα υποκινηθεί, διότι ξέρετε ότι για τα ανθρώπινα φάρμακα ε, υπάρχει πρόθεση της αρχικής, της βασικής έρευνας, αυτά που χρειάζονται για να υπάρχει μια αγορά, ε, εμπορία ουσιαστικά, όχι ένα νέο φάρμακο που θα είναι σε σχέση με κάποιο παλιό. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κερδοσκοπία για την βασική, την πρώτο επίπεδο έρευνα. Πρέπει να αποφύγουμε την συγκέντρωση ε, τη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια ορισμένων μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών που θα πάρουν την, ε, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στα κτηνιατρικά όπως έχει γίνει και με τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν το δίπλωμα τεχνίας για να ασκήσουν αυτήν την ε, δύναμη που έχουν και βεβαίω να κρατήσουν για τα χέρια του την αγορά. Εδώ λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε τις στρεβλώσεις που υπάρχουν για τον τομέα τη ανθρώπινη υγεία να τι αντιμετωπίσουμε τον προτέρων. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Πεντιτσίνη. Και τώρα τα μέλη της Επιτροπής. Μπορείτε να συνεισφέρετε στη συζήτηση. Έχουμε έξι συναδέλφους που έχουν ζητήσει χρόνο ομιλίας. Εάν υπάρχει κάποιος ακόμη, παρακαλώ να μας το πείτε τώρα. Αλλιώς κλείνει εδώ ο κατάλογος των αγορητών. Να αρχίσουμε με τον κύριο Λίζε. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή και όλους που συνεργάστηκαν για την Επιτροπή και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Τόνιο Μπόρκ ε, της προηγούμενης θητείας που υπέβαλε την πρόταση. Όταν η πρόταση αυτή υποβλήθηκε ήταν η ίδια μέρα που ο Ζωάν Κλοντ παρουσίασε την Νέα Επιτροπή. Κρίμα, γιατί είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχολεί για το θέμα τα υγείας. Γιατί φυσικά τα φάρμακα είναι από πλευρά δημόσιας υγείας το σημαντικότερο θέμα. Ευχαριστώ την ε, κυρία Γκόστετ για την εργασία που έχει ήδη κάνει για αυτό το θέμα και νομίζω ότι πρότεινε μερικές αναγκαίες βελτιώσεις. Είναι καλή βάση αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχει δίκιο η κυρία Γκροστέτ, πρέπει να τη βελτιώσουμε. Υποστηρίζω το στόχο να υπάρξει ε, πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και για τα κτηνιατρικά. Ένα πρώτο λοιπόν ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά και θα πω και εγώ κάτι γι' αυτό. Λέμε πολλά για τα αντιβιωτικά, αλλά θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν Ποια άλλα σημαντικά κτηνιατρικά φάρμακα υπάρχουν για τα ζώα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυτή την πρόταση και πού υπάρχουν ε, κάποιες ανησυχίες για αυτές τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων. Τώρα κάτι για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Σωστό είναι αυτό που λέει ο κύριος Χόσλινγκ. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα μέσω εκτιμήσεων του Οργανισμού Υγείας και του OECD, του ΟΣΑ, θεωρούμε ότι 25.000 ε, θανάτους κάθε χρόνο λόγω αντίστασης στα αντιβιωτικά. Και ίσως να είναι υψηλότερος αριθμός, όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ και ο συνάδελφος Φέντερλε από την Άγκρη. Και εγώ ίδιος συμμετείχαμε σε μια συζήτηση ένα μεσημέρι που είπαμε ότι μπορεί να είναι υψηλότερος αυτός ο αριθμός και πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι 25.000 θάνατοι δεν οφείλονται κυρίως σε κατάχρηση κτηνιατρικών αντιβιωτικών. Είναι κυρίως ε, λίγο κατάχρησης ε, αντιβιωτικών για ανθρώπους. Αλλά έχουμε προβλήματα στη γεωργία. Έχουμε μελέτες που λένε ότι για τα πουλερικά 90% των πουλερικών κατά τη σύντομη ζωή, ζωή τους, 35-40 μέρες, παχύνονται κατά 35-40 μέρε 90% παίρνουν αντιβιωτικά. Φανταστείτε τι θα σήμαινε. Εδώ είμαστε γύρω στα 100 άτομα. Εάν τι τελευταιε 35 35-40 μέρε είχε 90% εξημών πάρει αντιβιωτικά θα θεωρούσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό είναι καλό αυτό που εισάγει η Κομισιόν, 12 μέτρα για τη βελτίωση της χρήσης αντιβιωτικών, τα υποστηρίζω όλα και συμφωνώ επίσης με την Φρανσουάζ ότι πρέπει να δώσουμε καλύτερους ορισμούς. Με ανησυχεί βεβαίω αυτό το θέμα των αντιβιωτικών ε, τελευταίας γραμμής αμήνης. Και αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ περιορισμένο τρόπο για τα ζώα. Και η Κομισιόν λέει ότι πρέπει μέσω μιας καταξιοδότησης πράξης να το ορίσουμε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται, αλλά το θέμα αυτό πρέπει να μας απασχολήσει εμάς. Πρέπει εμείς να πούμε ποια αντιβιωτικά θα πρέπει να απαγορευτούν για τα ζώα, ποια πρέπει να χρησιμοποιούνται με περιορισμένο τρόπο και τι περιορισμούς θα εισαγάγουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν θα καταρτήσουμε ένα κατάλογο, αλλά να μας πει συγκεκριμένη κομισιόν τι θα κάνει. Και δύο άλλε ερωτήσει προς την Κομισιόν. Πρώτον, επί τη αρμόδια είναι η Άγκρη και εμεί θα κάνουμε μια γνωμοδότηση για τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τις ζωοτροφές. Και τέθηκε το ερώτημα, γιατί χρειαζόμαστε φάρμακα για τις ζωοτροφές. Έχει έννοια να βάζουμε αντιβιωτικά στις ζωοτροφές και αν το κάνουμε πρέπει να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένα. Γιατί χρειάζεται να τα βάζουμε στα, ε, στις ζωοτροφές. Θα μπορούσαμε να τα βάζουμε στο νερό που τους δίνουμε. Και κάποιο ε, ερώτημα είναι ευρύτερο αλλά πρέπει να το θέσουμε. Πέρα τα προβλήματα που έχουμε στον τομέα αυτό, το κύριο πρόβλημά μας είναι τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Γιατί να μην έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για να αποφύγουμε την αντίσταση στα αντιβιωτικά και για τους ανθρώπους. Έχουμε εδώ μια πρόταση, την έκθεση Grosstet, που βασίζεται στο άρθρο 14 και το άρθρο 168. Είναι εσωτερική αγορά και υγεία. Αυτή η νομική βάση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για τα φάρμακα για τους ανθρώπους οι γεωργοί έχουν δίκιο που λένε γιατί εμείς πρέπει να δώσουμε όλη αυτή την πληροφόρηση ενώ και στα ανθρώπια φάρμακα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα άρθρα, τα οποία δεν ισχύουν μόνο για τα φάρμακα για τα ζώα, αλλά και για τα ανθρώπια. Να το σκεφτεί λοιπόν η Κομισιόν. Σήμερα το απόγευμα Έχουμε αυτή την εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ε, πολιτικής φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των αντιβιωτικών και να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε. Ήρθε τώρα. Θα ήθελα τρία λεπτά ο καθένας σας. Ελπίζω να το δέχεστε. Επόμενος ομιλητής Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα χρησιμοποιήσω καν τρία λεπτά, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στην αντίσταση στα αντιβιωτικά. Η Μέριτ Πόλσεν ήδη ρώτησε γι' αυτό. Ρωτάω λοιπόν κι εγώ, γιατί οι κτηνίατροι να πουλούν τα ακτινατρικά φάρμακα τα οποία ήδη συνταγογράφουν. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα φάρμακα που παίρνουν οι άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι απλώς και μόνο θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να απαγορευτεί το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή το ότι έχουν το δικαίωμα οι κτηνίατροι να πουλούν και τα φάρμακα. Τα συνταγογράφουν, φτάνει. Ήδη το 1987 εμείς το έχουμε κάνει στη Δανία αυτό. Και όλος παραδόξος, το λέω βέβαια, μειώθηκε η κατανάλωση εκτινετρικών φαρμάκων. Φυσικά και υπάρχει σχέση ανάμεσα στον εγκαταλό. Όταν υπάρχει οικονομικό κίνητρο, ε, τι να κάνουμε, μπαίνουμε στον πειρασμό. Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Δεν λέω ότι πρέπει βέβαια να κάνουμε τους κτηνιάτρους να κερδίζουν πολύ λιγότερα, αλλά να βρούμε άλλους τρόπους να κερδίζουν αξιοπρεπώς τη ζωή τους οι κτηνίατροι. Γιατί πρόκειται εδώ πέρα και για την προστασία των ζώων, αλλά πρόκειται και για την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πιο αυστηροί. Αυτή λοιπόν θα είναι μια τροπολογία που θα υποβάλω. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σχερεμπέρικ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, έχω μερικές ερωτήσεις και εγώ όσον αφορά τα αντιβιωτικά και την αντίσταση στα αντιβιωτικά και πώς χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά για να αντιμετωπίσουν ασθένειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν την άκουσα καλά, λέει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά εξαίρεση κάποια αντιβιωτικά για τα ζώα και ότι θα απαγορευτούν ορισμένοι. Η ερώτηση όμω είναι πώ θα κάνετε αυτή τη διάκριση. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σα. Δεύτερον, πώ βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χρήση των μειοπαθητικών ε, μέσων ω φάρμακα σε σχέση με την πρακτική που ακολουθούμε εμεί στην Ολλανδία. Και τέλο, όσον αφορά τη χρήση πάντα των αντιβιωτικών, νομίζω ότι εδώ πέρα μιλάμε για λάθος χρήση τι σημαίνει όμως αυτό, πώς το καθορίζει αυτό, ποια είναι η λάθος ή μη λάθος χρήση των αντιβιωτικών, πώς καθορίζεται αυτή. Εγώ για χρόνια έχω ασχοληθεί με τους γεωργούς, με τους κτηνοτρόφους στη χώρα μου και είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που έχουν να είναι συγκεκριμένες. Θέλουμε τη σωστή ισορροπία. Θέλουμε υγιείς ανθρώπους, αλλά θέλουμε και υγιή ζώα και βέβαια και καλές ζωοτροφές. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ριβάζη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να περάσω ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να της πω ότι απλοποίηση δεν σημαίνει απορρίθμιση. Διότι όταν μιλάμε για διαθεσιμότητα τέτοιων προϊόντων, τι λέμε. Λείπουν φάρμακα, λέμε, και πρέπει να βρούμε περισσότερα φάρμακα για να αντιμετωπιστεί κάποια ασθένεια στα ζώα ή λέμε φάρμακα τα οποία να είναι σε τέτοιες τιμές ώστε οι κτηνίατροι, αν και εμείς προτιμάμε οι φαρμακοποιοί να χρησιμοποιούν. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια επίσης στις κλινικές δοκιμές. Μιλάμε για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Τι ακριβώς εννοούμε. Τι γίνεται με το Σολομό, ο οποίος εκτρέφεται και υπάρχει κάποιο είδους ψήλος ε, στον ε, Σολομό, ο οποίος τον καταστρέφει ολόκληρο. Χρειάζεται λοιπόν ένα φάρμακο, τον οποίο απαγορεύεται στην ε, ξηρά. Τι συνέπειες έχει. Υπάρχει μελέτη νομίζετε για τη σχέση ζώων ανθρώπων με τα λόγα. Τους δίνουμε αντιφλεγμονώδη και είδαμε ότι είχαμε σκάνδαλο και λέμε, α, προσοχή δεν πρέπει να το τρώμε αυτό το κρέας, γιατί τα αντιφλεγμονώδια αυτά επηρεάζουν και την υγεία των ανθρώπων. Λοιπόν, όταν μιλάτε για τη φαρμακοπαγρύπνηση στα ζώα, να ξέρετε ότι είμαστε στο στάδιο 0. Λέτε απλοποίηση. Ναι, αλλά η φαρμακοπαγρύπνηση πρέπει να αυξηθεί, να ενισχυθεί. Έπειτα, μας μιλάτε για καινοτομία. Τι μας προσφέρετε για την καινοτομία? Τα ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταλήγουν σε μονοπόλια σε διάφορες ονοκευτικές εταιρείες. Το έλεγε και συνάδελφος από τη ΕΣΥΑΡ νωρίτερα ότι ίσως πρέπει να βρούμε άλλα συστήματα ε, σχέσεις ιδιωτικού δημοσίου. Να υπάρχει καινοτομία με τα φάρμακα, αλλά να υπάρχει και διάθεση και όχι μόνο διπλώματα ευρεσιτεχνία. Συνθήκε πώληση τώρα. Η Δανέζα συνάδελφος μας το είπε πολύ καλά. Πώς θέλετε κτηνίατροι να κάνουν τη διάγνωση και οι ίδιοι να δίνουν τα φάρμακα εδώ πέρα. προφανώ και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αν ο κτηνίατρος που είναι κάποιο που δεν τον αφισβητώ, αλλά αν δεν δώσει αντιβιωτικά προφυλακτικά, ε, ο κτηνίατρο θα πάρει κάποιον άλλον. Ε, ο κτηνοτρόφο νόμου θα πάρει κάποιον άλλο κτηνίατρο που θα δώσει τέτοια φάρμακα. Και εδώ συμφωνώ με τη συνάδελφο Γκροστέτ. Δεν μπορούμε να λέμε συγχρόνω ότι θα μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών και συγχρόνω να λέμε ότι θα τα πουλάμε online ό,τι προσπάθεια θα κάνετε από τη μια μεριά, οι άνθρωποι θα πάνε και θα τα αγοράσουν μέσω του διαδικτύου. Έπειτα, αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αντίστασης ε, στα αντιβιωτικά. Ο συνάδελφος Λίζη έλεγε, μα δεν έχει και τόσο πολύ σχέση με τις εκτροφές. Μα όχι, ό,τι βρίσκουμε στο κρέας των ζώων, είτε στα βοηδή, είτε στα κουνέλια, οτιδήποτε, υπάρχει εντατική χρήση των αντιβιωτικών. Και αυτή η χρήση δημιουργεί βακτηρίδια τα οποία αντιστέκονται στα αντιβιωτικά στη συνέχεια και τα έχουμε παντού στις ε, κτηνιατρικές μονάδες. Μιλάμε για την φαγοθεραπεία. Μα αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η χρήση δηλαδή του στοιχείου εκείνου το οποίο θα καταστρέψει τα μικρόβια χωρίς αντιβιωτικά. Κύριε Γκροστέτ, τώρα όταν λέτε ότι θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιούμε τη δραστική ουσία. Μα οι πρώτες μελέτες για τα σκάνδαλα με τα ιστραγόνα ε, που γίνονται τελικά τα ψάρια κτλ. Τις ξέρουμε. Είδαμε ότι αλλάζουν τα οικοσυστήματα. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται μελέτες αντικτύπου. Και η δραστική ουσία συχνά ε, πρέπει να δούμε ποια ακριβώ είναι. Συνεπώς πρέπει να ενισχυθούν οι μελέτες αντικτύπου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενος. Ο μιλητής ο κύριος Φλόρενς. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα, αλλά άκουσα ορισμένου που μου έκαναν να σηκωθούν οι τρίχες. Εγώ είμαι Γιώργος και 28 χρόνια έχω ασχοληθεί πολύ με το χείριο κρέας. Και δεν έχω καμία αντίρρηση στο ότι υπάρχει υπερβολική χρήση αντιβιωτικών. Αλλά ακούω ορισμένου που λένε ότι δεν θέλουν να καταλάβουν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ discount στη Γερμανία και διαπιστώσετε ότι μπορεί να αγοράσει κανείς ένα ολόκληρο κοτόπουλο για 2,99 ευρώ, θα πρέπει να σκεφτείτε Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Ξεκίνησα πριν από πολλά χρόνια με 100 ε, χείρους και κατέληξα μετά από αρκετά χρόνια να έχω μια εκμετάλλευση χιλίων χείρων και αυτά δεν τα έκανα για να γίνω πλούσιος. Χρειαζόμουν χίλιους χείρους για να μπορέσω να θρέψω την οικογένειά μου γιατί οι τιμές πέφτουν τόσο πολύ. Σήμερα χρειάζεται κανείς 4.000 ζώα για να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με ένα-δυο παιδιά. Και αυτό είναι που οθεί τους ε, γεωργούς στη μαζική παραγωγή. Δεν το θέλουν οι ίδιοι. Ρωτήστε τους Ολλανδούς αδελφούς που έχουν στενή σχέση με τις τράπεζές τους. Γιατί είναι όλοι υπερχρεωμένοι. Και οι Γερμανοί το ίδιο. Άρα πρέπει να είμαστε λιγάκι προπροσεκτικοί. Και να θέσουμε το θέμα μιας λογικής, μιας δίκαιας, μιας σωστής τιμής. Όσον αφορά τη μείωση των αντιβιωτικών. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε ο Φρανσουάζ και ο Πίτερ Λίζε. Αλλά να κλείσουμε την πόρτα και να πούμε όλες αυτές τις ιδέες τις απαγορεύουμε. Είναι απλοϊκό. Κυρίως πρέπει να δούμε γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα αντιβιωτικά. Και εδώ φτάνουμε σε αυτό. Εάν έχεις 5.000 γουρούνια το χρόνο, θέλεις κάθε εβδομάδα 50 καινούρια που έρχονται από πέντε διαφορετικούς προμηθευτές και τότε αρχίζουν να αρρωσταίνουν γιατί έχουν όλα τα διαφορετικά μικρόβια, τα βάζεις ε, μέσα σε ένα υπόστεγο και τότε αρρωσταίνουν όλα. Και τότε κύριε Λίζε πρέπει να καταλάβετε γιατί πρέπει να το βάλουμε και στις ζωοτροφές. Άρα το θέμα είναι να υπάρξει εκπαίδευση για τις μορφές κτηνοτροφίας. Και ξέρω ότι η γεωργοί μου και εκτινοτρόφιμου, είναι απογοητευμένοι. Αν πρέπει όλα τα ζώα να είναι μέσα σε ένα υπόστεγο, ε, έχεις το πρόβλημα ότι έχεις πολύ διαφορετικά ε, μικρόβια. Χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων, συστήματα κατάρτισης, τα σωστά συστήματα εκτροφής Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε υπό τις συνθήκες που έχουμε οι γεωργοί μας να παράγουν ε, τρόφιμα που είναι κατάλληλα για να τα φάμε. Ευχαριστούμε. Τελευταίος μας ομιλητής, ο κύριος Άνιε. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω. Προφανώς ο υπεύθυνος απαντήσει θα είναι ο πρόσωπος της Επιτροπής. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τις ζωοτροφές και τα φάρμακα. Που μπορεί να περιλαμβάνουν δηλαδή φάρμακα. Ξέρετε ότι ετοιμάζει, συντάσει μια γνωμοδότηση η Επιτροπή μας από τη στιγμή για τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ζωοτροφές με φάρμακο. Εδώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ του θέματος που τώρα συζητάμε και του θέματος των φαρμακευτικών ζωοτροφών που θα έρθει επιτάπητο το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Ε, η ερώτηση είναι τι συσχετισμό βρίσκει η Επιτροπή μεταξύ των δύο θεμάτων και κατά πόσον είστε πρόθυμοι να δημιουργήσετε ένα κοινό πεδίο για να εξεταστούν από κοινό αυτά τα δύο ζητήματα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι κάπως πιο γενική. Αυτή τη στιγμή προβλέπουμε κάποιο είδου νομοθέτημα πλαίσιο. Και σχετίζεται με την ε, ευρωπαϊκή αγορά στο σύνολό της. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις για την διεκτατική εταιρική σχέση, τη TIP, από την σκοπιά του διεθνούς εμπορίου, κυρίως μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Και πώς βλέπετε την προοπτική να καλυφθεί και αυτό το θέμα στις συνομιλίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ζήτησε το λόγο και η κυρία Κάντεμπαχ. Μετά αυτά που είπε ο συνάδελφος Φλωρέντς, Θέλω να αντιδράσω. Γιατί εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονό ότι μιλάει ξέροντας περί πρόκειται. Και αυτά που είπαμε μου δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτή η αδειοδότηση με αυτή την εύκολη πρόσβαση στα αντιβιωτικά δηλαδή το ότι αυτό ο οποίο θα συνταγογραφεί τα πουλάει κιόλα, κιόλας και ότι επίσης μπορούν να πολιθούν και από το ίντερνετ σημαίνει ότι ποτέ δεν θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Και άρα θα τα έχουμε και στα τρόφιμά μας. Και οποιοδήποτε έχει άλλη τακτική δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Συμβάλλουμε λοιπόν. Ενισχύουμε στην πραγματικότητα το πρόβλημα. Γιατί διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Αντί να την απαγορεύουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάντεμπαχ. Και τώρα να πάμε πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να αντιδράσετε στις, απαντήσεις της στις που σας θέθηκαν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την ενδιαφέρουσα συζήτηση Θα προσπαθήσω να τη σωματοποιήσω για να καλύψω στο δυνατόν περισσότερο από τις ερωτήσεις και τα ζητήματα. Σε πολλές παρεμβάσεις θέσατε το θέμα των αντιβιωτικών, της προφυλακτικής χρήσης και της χρήσης αντιβιωτικών για λόγους προφύλαξης. Στην πρότασή μας Υπάρχει μια σειρά από διατάξεις για τα αντιβιωτικά. Μελετήσαμε όλους τους είδους πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να βρούμε την καλύτερη προσέγγιση. Και να δούμε πώς το προσεγγίζουν το θέμα αυτό τα διάφορα κάτι μέλη. Λόγω χάρη στη Δανία Έχουμε μια περίπτωση από τις καλύτερες. Δηλαδή η πολύ συστηματική ε, προσέγγιση με μεγάλη προσοχή ε, οδήγησε στην περιορισμό της χρήσης των αντιβιωτικών. Αλλά εδώ πρέπει να συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια όλοι οι φορείς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Από τους ίδιους τους κτηνίατρους που συνταγογραφούν μέχρι τους κτηνοτρόφους την ε, βιομηχανία και τις εταιρείε, τις δημόσιες αρχές κλπ. Πιστεύουμε ότι οι διατάξεις που προτείνουμε εξαρτάται πώς θα το ερμηνεύσετε, μπορεί να τις πείτε 12 ή 15 στην πρόταση. Είναι αρκετά περιοριστικές. Αλλά περιθώριο για νέες ιδέες υπάρχει και για βελτιώσεις. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά που το θέμα αυτό τίθεται και περιλαμβάνεται σε ένα κανονισμό. Ο δόκτωρ Λίζα ρώτησε εάν αυτό θα μπορούσε να καλύπτει κατά φάρμακα για ανθρώπους. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείναμε ένα πρόγραμμα δάσης για την μικροβιακή αντοχή. Προβλέπεται μια σειρά από δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για την ανθρώπινη, τη δημόσια υγεία. Άλλωστε προτείνουμε μια ρυθμιστική προσέγγιση που είναι αρκετά μοναδική. Οπότε το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε κιόλα όλα αυτά. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις για τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε τους κτηνιάτρους ως επαγγελματικό κλάδο και ως επαγγελματίες που ασχολούνται με την αγωγή και την προφύλαξη της ευζοίας των ε, ζώων. Ε, λεπτά ζητήματα, ξεκινώντας από την ερώτηση του κυρίου Κλέβα. Ε, το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους και την ανθρώπινη υγεία. Στα κράτη-μέλη δεν έχουμε ένα και μόνο σύστημα. Δεν είναι μόνο οι κτηνίατροι υπεύθυνοι για την ευζοία των ζώων, για την καλή του υγεία. Υπάρχουν και άλλοι επαγγελματίε εδώ. Γι' αυτό και πρέπει να το θυμόμαστε. Και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι εμπλέκονται. Και ασχολούνται με την ε, προστασία τη υγεία των ζώων. Πρέπει να προσέξουμε τον ορισμό μα. Στα περισσότερα βέβαια κατημέρια οι κτηνίατροι έχουν αυτή την αμοδιότητα. Σημαντικές ερωτήσεις τώρα. Τα επαγγέλματα που καλύπτονται και το πώς εργάζονται. Ξεκινώντας από τι ρυθμίσεις επιβάλλουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευσή τους, για την κατάρτισή τους, αλλά και τον τρόπο που μπορεί να πολλούν ή να περιορίζονται λόγω των ρυθμίσεων των κατών μελών. Συχνά, λόγω της διαθεσιμότητας των φαρμάκων, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει ο κτηνέτρος να πουλήσει αν δεν το έχει στη διάθεσή του στο ιατρείο του. Οπότε μπορεί το κάτω να αποφασίσει διαφορετικούς τρόπους πώλησης των φαρμάκων στα ζώα, για τα ζώα. Αλλά αυτό πρέπει να το δουν τα κράτη-μέλη. Είναι ένα σημαντικό σημείο. Στην ανθρώπινη υγεία κάποια κράτη-μέλη επιτρέπουν κάποια φάρμακα αλλά είναι εξαίρεση και είναι, αφορά μόνο την ε, ανθρώπινη υγεία. Για το θέμα της καινοτομίας έχουμε διπλή προσέγγιση μάλλον δύο διαφορετικές, η κυρία Γκροστέτ είπε, ότι δεν είμαστε ίσως αρκετά φιλόδοξοι για να προωθήσουμε την καινοτομία και να, πρέπει να βρούμε και άλλες πρωτοβουλίες για να φτάσουν νέα προϊόντα ως την αγορά. Ο κύριος Πλέβα είπε ότι πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και τιμών. Θα φροντίσουμε κάτι να συμπεριληφθεί στην πρόταση για να μπορέσουν ε, οι ερευνητέ των φαρμακοβιομηχανιών ή γενικότερα όσοι προτείνουν νέα φάρμακα και προϊόντα να φτάσουν στην αγορά. Γενώσιμα. Ε, ενδιαφέρουν πάντα την αγορά, αλλά το θέμα είναι να βρούμε και το σωστό ρυθμό για τα εντελώς νέα προϊόντα. Οι τιμές δεν σχετίζονται απαραίτητα με το επίπεδο προστασία στο IPR, αλλά με τι μελέτε αντεκτύπου. Οι κανόνε του IPR είναι οι ίδιοι για όλου σήμερα. Ίσως χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για να μπορέσουν να φτάσουν στην αγορά τα προϊόντα σε καλύτερε τιμέ. Και τώρα να έρθω στις ε, πωλήσει στο ίντερνετ. Οι διατάξεις που εγκρίναμε για τα, ανθρώπινα, για τα φάρμακα για την ανθρώπινη κατανάλωση με την σχετική οδηγία του 2011 διασφαλίζει ότι όσοι πολλούν στο διαδίκτυο ε, ελέγχονται από τις εθνικές αρχές ε, στη χώρα εγκατάστασης. Δεν μπορεί και λοιπόν κανείς να πουλάει στο διαδίκτυο χωρίς κανέναν έλεγχο. Ελέγχονται από τις εθνικές αρχές όλοι αυτοί. Η ερώτηση είναι αυτό πώς θα συνδυαστεί με τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και τι είδους περιορισμούς μπορεί να έχουμε στις πωλήσει. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη συζήτησή μας και να είμαστε βέβαιοι ότι η διαθεσιμότητα των ε, φαρμάκων για πολλούς θα είναι το βασικό κίνητρο και κινητοποίησε και όλοι μας την πρόταση. Πιστεύουμε επίσης, εφόσον μιλάμε για τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες εξελίξεις στον χώρο των πωλήσεων στο διαδίκτυο. Μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά η πώληση φαρμάκων. Μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρονικές συνταγές σε πολλα κάτι κράτη-μέλη. Και εκεί ηλεκτρονικά φαρμακεία. Η συλλογή δεδομένων ηλεκτρονικά στο μέλλον. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές για την αγορά θα αρχίσουν να υλοποιούνται τα ερχόμενα χρόνια, οπότε θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Επειδή δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, να επικεντρωθώ ακόμη σε κάτι που τέθηκε από την κυρία Γκροστέτ για τις κλινικές δοκιμές για την ε, παραγωγή ζωοτροφή στα ζώα που χρησιμοποιούνται μάλλον που, από τα οποία παράγονται και τρόφιμα. Εδώ η περίοδος απόσυρσης πρέπει να έχει πολύ σαφή όρια. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε σίγουρα. και πώς αυτό σχετίζεται με τις φαρμακευτικές ζωοτροφές και την ε, σχετική πρόταση. Συνεργαζόμαστε στενά. Συμπεριλαμβανόταν αυτό στην δέσμη μέτρων. Προσπαθούμε να μην υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ των δύο προτάσεων. Η Επιτροπή Άγκρη είναι υπεύθυνη για αυτήν την συζήτηση, αλλά και εμεί στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο συστημάτων. Ίσως να ολοκληρώσω με τα θέματα της φαρμακοεπαγρύπνησης και πώς αυτό το νέο σύστημα μπορεί να αποδώσει περισσότερα. Χάρη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, από τον Ιανουάριο του 2000 είχαμε Ιανουάριο του 2000, το παραλαμβάνω, είχαμε 1123, 1123 εκθέσεις που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια φαρμακών και διαρκώς επικαιροποιούνται ως σήμερα. Μόνο 3,3% οδήγησαν σε αιτήματα για αλλαγή στις πληροφορίες περί του προϊόντος. Δηλαδή το 97% σχεδόν δεν είχαν κανένα, καμία αρνητική ένδειξη. Τώρα στο νέο σύστημα θα έχουμε ακόμα ευρύτερη συγκέντρωση πληροφοριών. Ηλεκτρονική υποβολή, σήμανση. Το θέμα δεν είναι πόσες εκθέσεις οι σημάνσεις θα λάβουμε, αλλά ποια είναι η, αξία, το κύρος των εκθέσεων αυτών για τη λήψη των αποφασιών μας. Νομίζω το νέο σύστημα θα μειώσει το άχθος, αλλά ταυτόχρονα θα πετύχει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο πρόεδρος μου κάνει νοήματα ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ. Και στη διάθεσή σας για την παρουσίαση της δεύτερης πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε έτσι αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση με τόσο τεχνικά στοιχεία. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, υπενθυμίζω τροπολογίες προκειμένου να μεταφραστούν και τα... Α, μια στιγμή. Η κυρία Γκροστέτ, η συγγετριά μας, θέλει να αντιδράσει μετά από τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις παρατηρήσεις των μελών. Πριν Λοιπόν, σας δώσω αυτές τις τεχνικές πληροφορίες για προθεσμίες, κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομη, γιατί αφιερώσαμε πράγματι πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το ζήτημα, που είναι όμως και σημαντικό. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ακούγοντάς τους, διαπιστώνω ότι προβληματιζόμαστε για πάρα πολλά σημεία και οι προβληματισμοί μας συγκλίνουν ουσιαστικά. Είμαι πεπισμένη ότι με συνεργασία θα καταλήξουμε σε ένα βελτιωμένο κείμενο και ελπίζω θα πηγαίνει πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, χοντρικά, θα αναφέρω κάποια σημεία στο οποίο αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι χωρίς να τους κατανομάζω. Ναι, όσον αφορά την σήμανση και τη συσκευασία. Είναι αλήθεια αυτά που είπατε. Και όσον αφορά το φαινόμενο αυτό χιονοστιβάδας, όντως η χρήση των φαρμάκων αυτών στην κτηνιατρική πρέπει να γίνεται αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Να είμαστε πολύ απαιτητικοί. Έρχομαι τώρα στο θέμα της καινοτομίας και της τιμής των προϊόντων. Πράγματι πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Υπάρχουν προβλήματα, τα ανέφερε και πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά. Εγώ έχω επιλέξει να μην πάω τόσο μακριά όσο λέει η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άκουσα όμως και τους συναδέρφους και μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για τα γενώσιμα είναι να τα δούμε μακροπρόθεσμα. Και νομίζω ότι η προστασία της καινοτομίας είναι υπέρ τους τελικά. Για τη συνταγογράφηση υπήρξε μια ερώτηση. Ναι, θα υπάρξει ένα μοντέλο για τις ε, συνταγογραφήσεις αυτές. Το άρθρο 110 αναφέρει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφέρονται σε κάθε συνταγή. Θα έχουμε δηλαδή ένα αρμονισμένο έγγραφο για αυτό το σκοπό. Όσον αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών μεταφυλακτικά, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ε, υπάρχει, εκδηλωθεί μια ασθένεια και χρειάζεται αντιβιωτικό, πρέπει να θεραπεύσουμε, μάλλον να αντιμετωπίσουμε το εδεχόμενο ε, μόλυνσης και των άλλων ζώων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια διάγνωση συγκεκριμένη και να αποφεύγουμε τη χρήση των αντιβιωτικών αν δεν υπάρχει πραγματικά λόγος για να χρησιμοποιηθούν. Επίσης θα έλεγα στον σκιώδη συγγετή από το FDD που κατηγορεί την πρόταση γιατί λέει ότι είναι πολύ υπέρ της βιομηχανίας και ότι δεν στοχεύει κυρίω τη δημόσια υγεία. Σας διαβεβαιώ αγαπητέ συνάδελφε, το μόνο που με απασχολεί εμένα είναι η υγεία των ζώων και οι συνέπειες της βέβαια και επί της υγείας των ανθρώπων είναι αλληλένδετα. Ισχύει και για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Έχουμε τη σπάθα του απάνω μας. Είναι η αντίσταση στα μικρόβια και στα αντιβιωτικά στη συνέχεια. Γι' αυτό και πρέπει να πιέσουμε την φαρμακευτική βιομηχανία να κάνει έρευνα για νέα φάρμακα. Ακόμα και αν θέλουμε τα νέα αυτά αντιβιωτικά να χρησιμοποιούνται πολύ περιορισμένα και να τα ελέγχουμε. Παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη για καινοτομία στα φάρμακα. Δεν είναι σε αντίθεση αυτά τα δύο μεταξύ τους. Πρέπει να βελτιώσουμε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Δείτε τι γίνεται με τις μέλισσες. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην εξαφανιστούν οι μέλισσες. Και αντίθετα πρέπει να φροντίσουμε να πολλαπλασιαστούν, να έχουμε περισσότερες μέλισσες στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε επαγγελματικά το θέμα των ε, παραγωγών μελιού. Αλλά πάντως είναι ένα πρόβλημα. Μα αναφέρθηκε και εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες. Όταν πετάμε αντιβιωτικά στο νερό για τα ψάρια, ε, βέβαια και υπάρχει πρόβλημα. Συνεπώς, όλα αυτά πρέπει να διαμετωπιστούν. Τώρα έχουμε στην πώληση στο διαδίκτυο. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Πιστεύω ότι η πώληση αντιβιωτικών ή άλλων φαρμάκων στο διαδίκτυο πρέπει να απαγορεύεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακόμα και αν δεν θέλω εδώ να τα βάλω με τους ε, κτηνοτρόφους, αλλά είναι τόσο εύκολο να πάει κανείς σε κάποια ιστοσελίδα που δεν βρίσκεται που έλεγχο και να βρει αντιβιωτικά που να μην είναι καν αυθεντικά, να είναι πλαστά. Έτσι καλώ θα χρησιμοποιούμε τόσο συχνά τα αντιβιωτικά. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος για τέτοια φάρμακα που δεν ελέγχονται και μπορεί να είναι πλαστά ακριβώς. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μας λέει ότι θα είναι ένα σημείο διαφωνίας με το Συμβούλιο. Ναι, μα εδώ είμαστε για να προστατεύσουμε την υγεία. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ είναι υπέρ του να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με αυτό το ζήτημα. Θα συνεργαστώ λοιπόν μαζί σας, με όλους σας, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, πάντως σας ευχαριστώ όλους και Θέλω να συνεργαστώ με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και με όλους τους ευρωβουλευτές για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να είναι όσο γίνεται καλύτερο. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ωραία. Χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία. 13 Απριλίου πρέπει να πάει στη μετάφραση το κείμενο της εισηγήτριας. 6 και 7 Μαΐου θα το εξετάσουμε στην Επιτροπή μας. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 15 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα 15 Ιουνίου, 4 το απόγευμα. 4 μετά Μεσενδρίας. Θα ψηφίσουμε στις 22 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές δηλαδή, και δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πότε θα πάει στην Ολομέλεια. Περνάμε στο επόμενο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Έχει άμεση σχέση με αυτό που μόλις συζητήσαμε βέβαια. Πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού 726 κάθετος 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδεια και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για ακτινιατρική χρήση και για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Θα ακούσουμε εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη συνέχεια τον εισηγητή μας και τους σκιώδης. Περνάει ο χρόνος και έχουμε και αυτό το θέμα και άλλο ένα μετά να συζητήσουμε. Οπότε σας παρακαλώ να δεχτείτε κάποιο περιορισμό στο χρόνο ομιλίας. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνοψίσει παρακαλώ σε 8 λεπτά το πολύ τη θέση της Επιτροπής. Ο συγκριτής 5 λεπτά, 3 λεπτά ο καθεσκιώδης και αν υπάρξουν και άλλοι ευρωβουλευτές που θέλουν το λόγο, Δύο λεπτά καθένα. Έτσι καλώς πολλά από τα ζητήματα έχουν συζητηθεί με το προηγούμενο θέμα, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να τηρήσουμε το χρόνο μας για να έχουμε χρόνο και για το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι και το τελευταίο. Συνεπώς, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τροπολογίες ο κύριος Ρης. Ο κύριος Ρης θα παρουσιάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός είναι αυτόνομος. Και για να το επιτύχουμε αυτό αφαιρέσαμε από το κανονισμό 726 2004 όλες τις διατάξεις που αφορούν τα κτηνιατρικά και τα μεταφέραμε στο νέο κανονισμό και μετά την έναξη ισχύω της συνθήκης Λισαβόνας πρέπει να ε, ε χρησιμοποιήσουμε όρους Λισαβόνας Άρα όλες οι αναφορές ε, για επιτροπολογία μετατρέπονται σε αναφορές σε κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Να λοιπόν η δομή. Όλες οι διατάξεις. Στους τίτλους 1, 2, 3, 4, 1 και 5 και για τα παραρτήματα όλες αυτές οι διατάξεις περνάνε στο νέο κανονισμό. Προτείνουμε ο τίτλος 3 να καταργηθεί και να πάνε αλλού οι διατάξεις αυτές. Οπότε καταργήσαμε όλες τις αναφορές στα κτηνιατρικά και ε, στο κείμενο και στα παραρτήματα του κανονισμού 726. Για παράδειγμα, μετα, μετατρέπονται διάφορα άρθρα στη νέα διαδικασία αυτή που ανέφερα και το άρθρο 61 που αφορά τη διαδικασία των μελών της Επιτροπής για τα κτηνιατρικά φάρμακα όλα αυτά τροποποιήθηκαν. Τώρα, το κόστος περνάει στις κατευθυνότητες πράξεις για τα τέλη. Έτσι παίρνουν τις αποφάσεις. Εμείς προτείνουμε και το Συμβούλιο εγκρίνει στις διαχειριστικές επιτροπές. Στο νέο κανονισμό για τα τέλη για την φάρμακοεπαγρύπνηση έχουμε νέους κανόνες σε αυτό τον κανονισμό. Στο νέο αυτό κανονισμό 658 14. Τι θα ισχύσει λοιπόν, η πρόταση λέει ότι η Επιτροπή θα τροποποιεί μέσω εφαρμοστικών πράξεων τα τέλη αυτά υπό τον έλεγχο των κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Τα εθνικά τέλη λοιπόν δεν καθορίζονται με βάση την πρόταση αυτή γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις για την ε, δομή αυτών των τελών. Όλες αυτές οι αλλαγές μας επιτρέπουν μια ευανάγνωστη, διαφανή και ρωμαλαία πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο εισηγητής μας κύριος Τρανσέσκου έχει πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, είναι πολύ θετική αυτή η αποσύνδεση της έγκρισης ε, εμπορίας για τα κτηνιατρικά από τα ανθρώπια για να λάβουμε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου. Ωστόσο, το κείμενο πρέπει να λέει σαφώς ότι ο οργανισμός θα έχει το ρόλο του για την αδειοδότηση και την επίβλεψη ε, των ιατρικών μέσω της ε, συγκεντρωτικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε νέα αρμοδιότητα θα δοθεί στο φορέα φαρμάκων θα πρέπει να αναφερθεί κατά την ε, μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση του 726 και κάποια θέματα που αφορούν το προϋπολογισμό του οργανισμού φαρμάκων και τα τέλη που θα λαμβάνει χρειάζονται διευκρίνηση. Για παράδειγμα, το άρθρο 70 που είναι η νομική βάση για την πληρωμή οποιονδήποτε τελών στον οργανισμό φαρμάκων, είτε είναι ανθρώπινα, ανθρώπια, είτε εδρικά τα φάρμακα. Εκεί αναφέρεται λοιπόν πώς πρέπει να γίνεται. Αλλά ξέρουμε ότι θέλει να, αναθεωρήσει και το, να θεωρήσει και το 297 για το γενικό κανονισμό για τα τέλη προς τον οργανισμό φαρμάκων. Ο νέος κανονισμός, ο πρώτος, όμως προτείνει μια εκτελεστική, μάλλον μια εφαρμοστική πράξη. Άρα τι περιεχόμενο θα έχει η αναθεώρηση του κανονισμού για τα τέλη. Και πολύ περιορισμένος είναι ο ρόλος επίβλεψης του Κοινοβουλίου για μια εφαρμοστική πράξη. Ενώ εγώ θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στον καθορισμό των τελών προς τον οργανισμό φαρμάκων, όπως κάναμε και για τα τέλη για την φαρμακοεπαγρύπνηση πρόσφατα. Οπότε, παρακαλώ, να διευκρινίσετε περαιτέρω στο άρθρο 70 ποιο νομικό μέσο θα χρησιμοποιήσετε και πώς ε, προβλέπετε να αναθεωρήσετε τον κανονισμό για τα τέλη. Σε αυτή τη ε, νέα προσπάθεια, το νέο εγχείρημα καθορισμού των τελών θα συμμετάσχει πλήρως το Κοινοβούλιο. Ο κανονισμός για το γενικό καθεστώς τελών θα πρέπει να είναι η προσωρινή νομική βάση μέχρι να αρχίσει να ισχύει η νέα εφαρμοστική πράξη ή ο νέος κανονισμός και μόνο τότε μπορεί να ακυρωθεί η βασική πράξη. Η Κομισιόν θα πρέπει να δηλώσει σαφώς μέσω της πρότασης που έχουμε μπροστά μας τις προθέσεις της, ούτω ώστε ο οργανισμός φαρμάκων να μην ε, ε, ε, αντιμετωπίσει ασάφεια για το πώς θα ορίζονται και πώς θα πληρώνονται τα τέλη. Πρέπει λοιπόν να αρχίσει αρκετά νωρίς η προετοιμασία της, της πράξη ε, πράξης για να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε για την περίπτωση των ε, ανθρωπίων φαρμάκων στα πλαίσια της διαδικασίας φαρμακοεπαγρύπνησης. Το άρθρο 70 προτείνει η πράξη αυτή ότι θα είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε τέλη προς τον Οργανισμό Φαρμάκων για ανθρώπια ή κτηνιατρικά φάρμακα. Όμως, το πόσες εφαρμοστικές πράξεις θα επιλεγούν θα έχει επιπτώσεις στη δομή του προϋπολογισμού του οργανισμού. Και θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια κοινή δομή για τα τέλη. Διευκρινίστε λοιπόν παρακαλώ ως Επιτροπή εάν θα έχετε μία ή δύο εφαρμοστικές πράξεις. Και τελευταίο. παρατήρησα ότι η Κομισιό λέει ότι αυτή η νέα εφαρμοστική πράξη θα βασιστεί στο κόστος των κρατών μελών και του οργανισμού. Από πλευράς αρχής το καλωσορίζω. Αλλά θα πρέπει η Κομισιό να λάβει υπόψη τις διομορφίες του κλάδου και να διασφαλίσει ότι τα τέλη αυτά θα εξακολουθήσουν να είναι λογικά για τον κλάδο για να υπάρχουν τα αναγκαία κτηνιατρικά φάρμακα στη διάθεση του κλάδου. Μήπως θα είχε σχόλια εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που τηρήσατε το χρόνο ομιλίας. Τώρα περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτα απ' όλα οι σκιώδεις του, του ΕΛΚ, η κυρία Κωνστέτ και πάλι. Ναι, στην πραγματικότητα δεν είμαι εγώ ισχυώδης εισηγήτρια, αλλά εξ ονόματος του συναδέλφου Σύριο ε, παρεμβαίνω. Δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Όπως εξήγησε ο εισηγητής, το κείμενο αυτό έρχεται μαζί με το σχέδιο κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Πρόκειται για ένα κείμενο άκρο τεχνικό. που σκοπό έχει να εκφράσει με νομικό τρόπο τις επιπτώσεις που θα έχει η αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Αυτό λοιπόν που προέχει είναι να έχουμε μια μεγάλη να συμβαδίζουν μάλλον τα δύο κείμενα και να υπάρχει συνοχή. Ο συνάδελφός μου ο κ. Σύριο ε, δεν έχει εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα στην έκθεση αυτή. Δεν θα υπάρξει λοιπόν δυσκολία να ακολουθήσουμε την ε, γενικότερη θέση του εισηγητή. Αλλά είναι, όπως και εσείς το είπατε, είναι πολύ ε, ανήσυχος για το θέμα των τελών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως θέμα που θα πρέπει να στρέψουμε όλοι μας την προσοχή η αλλαγή της νομοθεσίας που θα επηρεάσει και τα κτηνιατρικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσει ένα επιπλέον ε, φόρτο εργασίας για τον οργανισμό φαρμάκων και αυτό ακόμα και με την πρόβλεψη κεντρικών διαδικασιών. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια αντιστάθμιση λοιπόν με τέλη που, ε, τον οποίο θα μας απασχολήσει το ποσό και το βάρος τους. Ε, για όσους θα πρέπει να τις καταβάλουν. Αυτά είναι τα βασικά σημεία επί των οποίων ο κύριος Σύριο ήθελε να επιμείνουμε. Το κάνω αυτό στη θέση του. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μείνω για τη συζήτηση. Με περιμένουν σε άλλη συνεδρίαση. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να ακολουθήσουμε την θέση του εισηγητή μας. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Μπίχα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα από τα ζητήματα που μας απασχολούσαν και με το προηγούμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ίσως να μιλήσουμε για την ε, συμμόρφωση, και το κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν ε, με τη συνθήκη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 3.1α ε, τον τρόπο που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Χαστοξουσιοδότησης πράξεις και τις προτάσεις τους με τα σχετικά δεδομένα. Ε, εδώ πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να του δώσουμε λιγότερη σημασία από ό,τι το αξίζει. Να βασιστούμε λοιπόν στο άρθρο 192. Δεν θα πρέπει να είναι μάλλον εφαρμοστική πράξη, αλλά εκτελεστική μάλλον πράξη, αλλά κατά εξουσιοδότηση πράξη. Με συγχωρείτε για τον μπέρδεμα. Αυτό είναι το τεχνικό ζήτημα. Τώρα για τα τέλη, αυτό είναι πραγματικά αμφιλεγόμενο. Θα επηρεάσει το πώς θα ερμηνεύσουμε το θέμα του γραφειοκρατικού άκτου. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αγορά, ε, αυτό που μας λένε είναι ότι φοβούνται ότι θα πληρώσει τα σπασμένα ο δικός τους κλάδος. Για το σύστημα διοδότησης τώρα, για τις άδειε, οι αποκεντρωμένες διαδικασίες ή οι απλουστευμένες εκδοχές τους δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν, μάλλον αυστηρότεροι πρέπει να γίνουμε, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της δημόσιας υγείας και για τις κυρώσεις. Δεν υπάρχουν πρόστιμα Εάν υπάρχει κάποιο φορέα που δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του, αλλά προβλέπει φάρμακα, δεν ξέρουμε τι κυρώσει θα υπάρχουν, τι είδου επιπτώσει, τι ευθύνε, ποιο θα το καλύψει και ούτω καθεξή. Και τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, έχουμε και τα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα. Είμαι γιατρός να σας πω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα φάρμακα που έχουν ε, επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μέσνερ που είναι σκιώδης εκ μέρους των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Πολλά έχουν ήδη υποθεί. Πολύ σωστό ότι θέλουμε να απλοποιήσουμε και να βάλουμε σε ένα κείμενο τις διατάξεις αυτές και βεβαίως για τις εφαρμοστικές πράξεις ε, το Κοινοβούλιο πάντα θέλει να εξετάσει αν είναι τεχνικό ή μήπως και πολιτικό το θέμα. Αυτό πρέπει να το δούμε πιο αναλυτικά στα πλαίσια ακριβώς ε, των συναντήσεων των σκιωδών. Οπότε θα πω ότι θα συζητήσω με τους συναδέλφους και θα υποβάλω τροπολογίες. Καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν θέλει να απλουστεύσει τη διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι επαρκώς ετυλογημένη η πρόταση, γιατί είναι θέμα υγείας ε, και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα φάνε τα ζώα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΟΕ, η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να παρέμβω τώρα. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε για την σύντομη παρέμβασή σας. Πράσινη, ο κύριος Χόσλιν. Συμφωνώ με τους προηγούμενους. Είναι πολύ τεχνική αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να ελέγξουμε εάν το Κοινοβούλιο συμμετέχει παρκώς γιατί έχουμε προβλήματα με τις εφαρμοστικές πράξεις. Το θέμα των τελών, βεβαίως έχουμε ακούσει επικρίσεις, δεν είναι απλό. Θα πρέπει να αποφύγουμε να φυγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντίθετα με προηγούμενους πρέπει να πω ότι δεν θα πρέπει επίσης ε, να τεθούν σε μειονεκτική θέση τα ομοιοπαστικά φάρμακα. Αυτά και κατά τη διαδικασία θα περάσουμε στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Νικόλα Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους και και τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Είναι άκρος τεχνικό, όπως υπόθηκε. Και διακρίνει εδώ τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από τα κτηνιατρικά φάρμακα. Συμφωνούμε και εμείς με αυτή την αποσύνδεση. Από την άλλη, είμαστε υπέρ της κατεξοδότησης πράξης που προβλέπουν δικαίωμα αναρρησικηρίας για τον νομοθέτη. Σε αυτό όμως το επίπεδο και μετά όπως υπόθηκαν και για το προηγούμενο θέμα, Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπορεί να προχωρήσει. Θα ε, για τι λεπτομέρειε με του υπόλοιπου συνεισηγητές. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλο το λόγο. Οπότε πάμε πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ρίσου για να προσπαθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις ή να κάνει ό,τι άλλες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. σε ευχαριστώ πολύ. Γενικά μιλώντας, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να εξετάσουμε τον, την πρόταση αυτή με την κύρια πρόταση που συζητήσαμε πριν όσον αφορά πρόστιμα κυρώσεις και άλλα. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτήν την πρόταση αυτή καθεαυτή είναι ρύθμιση τελών και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Γιατί η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει εφαρμοσμένες ε, διατάξεις αυτήν εδώ την πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του C427 εξέτασε πώς εφαρμόζονται και πώς ρυθμίζονται τα τέλη σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επρόκειτο για την ΕΚΑ, για παράδειγμα, για τα χημικά. Και το δικαστήριο πρότεινε ουσιαστικά αυτό το σύστημα, αυτό μας πρότεινε. Ξέρουμε ότι στη φαρμακοθρήμηση, για παράδειγμα, υπάρχουν άλλες επιλογές. Είναι αλήθεια ότι δουλεύουμε πάνω στην οργάνωση των τελών. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αλλά και τους εθνικούς. Υπάρχει λοιπόν το δίκτυο των οργανισμών και πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί καλά. Όπως θα θυμόσαστε από τις συζητήσεις για τα τέλη φαρμακοπαγρύπνησης ήταν δύσκολο γιατί είχαμε το εκτιμόμενο κόστος, το πιθανό κόστος Γι' αυτό λοιπόν εδώ θέλουμε να φροντίσουμε η πρόταση να συμφωνηθεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τους Εθνικούς Οργανισμούς Φαρμάκων. Φυσικά θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλά μπορεί να πάρει χρόνο. Και εμείς ακολουθούμε και τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξωτερική αξιολόγηση της πρότασης, κάτι το οποίο σχεδιάζουμε. Τώρα, για το κατά πόσο τα τέλη θα αλλάξουν την προσβασιμότητα, αυτό είναι καλό. Αυτό ακριβώ είναι και το θέμα μας, ότι θέλουμε να βρούμε ε, μια τέτοια διάρθρωση τελών που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μπαίνουν στο σύστημα, να μην το μπλοκάρουν. Εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς, από τη δυνατότητα κερδών που υπάρχει για τους ερευνητές. Φυσικά η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι είναι με τα ανθρώπινα φάρμακα για ανθρώπινη κατανάλωση. Αν χρειάζεστε τώρα διευκρινήσεις για το μεταβατικό στάδιο, ευχαρίστω. Δεν πρέπει να υπάρξει κενό. αν θέλετε να τα διευκρινίσουμε περισσότερο βεβαίως. Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 70, έτσι όπως προτείνεται τώρα, επιτρέπει την ε, καλή, πιστεύω, διάρθρωση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες φαρμάκων για ανθρώπινη και για ε, εκτενοτοφική κατανάλωση. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Τανασέσκο, εισηγητής, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διάφορα σημεία τα οποία ανέπτυξε. Χωρίς τις εξηγήσει ίσως να είχαμε μια δύσκολη συζήτηση. Για το θέμα της πολιτικής πτυχής και της τεχνικής πτυχής, εγώ θα έλεγα ότι το θέμα μας είναι η υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σας διαβεβαιώ, έτσι θα το αντιμετωπίσω. Με μεγάλο σεβασμό και σοβαρότητα. Τέλος, αλλά και λιγότερο σημαντικό, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστήσω και τους συναδέρφους, τους κοιόδες εισηγητές για τη βοήθειά τους και να σας διαβεβαιώσω για το ότι θα λάβω υπόψη μου κάθε πτυχή που αναφέρθηκε. Θα προσπαθήσω έτσι. Ελπίζω τουλάχιστον να έχω την καλύτερη δυνατόν έκθεση σε ευχαριστούμε πολύ. Χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. 15 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒ στις 22 Σεπτεμβρίου και θα αποφασιστεί κάποια στιγμή και πότε θα πάει στην Ολομέλεια. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλες σας τις παρεμβάσεις σε αυτή τη συζήτηση. Και θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα και που είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το σχέδιο Juncker δηλαδή. Θα ζητήσω τώρα από την συντάκτρια γνωμοδότησης, την κυρία Μίρια Μαντάλη, να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Και μετά θα ακούσουμε τους κοιόδης. Σύμφωνοι, παρακαλώ, κύριε Νταλή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήδη είχαμε κάποιες θερμές συζητήσει στην Ολομέλεια, την Επιτροπή Οικονομικών Προπολογισμών και σε άλλες επιτροπές των μεταφορών για αυτό το ειδικό και κατεπήγον θέμα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, όπω είπατε το πρόγραμμα Juncker. Πριν από λίγε εβδομάδε δηλάβαμε το σχέδιο πρόταση. Η βασική ιδέα του προγράμματο αυτού είναι να αξιοποιήσει τις ιδιωτικέ επενδύσει μαζικά ω ένα πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική ανόρθωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την οικονομική και κοινωνική συνοχή ε, και τους ε, περιβαλλοντικούς μας στόχους. Για την βιώσιμη και ε, απελαγμένη από τον άνθρακα και ε, πρόσφορες προς τη χρήση των πόρων πολιτική μας χρειάζεται αυτού του είδους η ανάπτυξη. Από τη σκοπιά μου και προ... του περάσω στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ να πω ότι με τους σκιώδεις προσπαθήσαμε να συμμεβάσουμε τις απόψεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων και να συμπεριλάβουμε τις προτεραιότητές τους στην ίδια την γνωμοδότηση. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους σκιώδεις για την συνεισφορά τους θα ήθελα να σταθώ σε επτά βασικά ζητήματα που από την σκοπιά της ΕΝΒΗ είναι ιδίω σημαντικά. Πρώτον, είναι σημαντικό η ΕΤΕ να δώσει προτεραιότητες και να στηρίξει βιώσιμα έργα με έμφαση στι ανανεώσιμε πηγέ και τι τεχνολογίε χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και βέβαια με ε, βάση του στόχου για τη βιώσιμη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2050 και το κλίμα. Δεύτερο σημείο. Μέσα από τη γνωμοδότηση, οι στόχοι να διευκρινιστούν κάποια θετικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι επενδύσει θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητε στι βιώσιμε μεταφορέ, στην προώθηση τη βιώσιμη κινητικότητα, στην ηλεκτροκίνηση και την ε, εκτεταμένη χρήση των ενεργειακών, των εναλλακτικών ενεργο, εν, πηγών ενέργεια, με του ηθεί μετρητέ ε, και του διασυνδέτε για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, την ε, ε, ενεργειακή ε, μετάβαση, βεβαίως και την στήριξη έργων ενεργικής αποδοτικότητας, ιδίως την ανακαίνιση από ενεργειακής πλευράς των κτηρίων. Πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν έργα που να πληρούν τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, τους στόχους της ανάκαμψης της οικονομίας, την βιώσιμη κινητικότητα και τους στόχους της μετάβασης της αγοράς. Χρειαζόμαστε οι επενδύσεις του ΕΦΣΥ να δίνουν ισχυρή στήριξη στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη τέτοιες επενδύσεις. Θα πρέπει να δίνουν περισσότερη προσοχή και στοχευμένες επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων ε, πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, για τη χαμηλή κατανάλωση και τεχνολογικές λύσεις που βρίσκονται ακόμη στην φάση της δοκιμής με την οικολογική καινοτομία και την ε, έρευνα για τα νέα καινοτόμα φάρμακα. Οι επενδύσεις που θα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική, Επενδυτική Στρατηγική μαζί με τους δημόσιους πόρους βάσει της γνωμοδότηση της ΕΝΒΗ θα πρέπει να περάσουν από μελέτη αντικτύπου, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βάσει των ενεργειακών στόχων, τη ε, ε, σωστής των πόρων και τη απαλλαγμένη από τον άνθρακα πολιτική μα. Πρέπει να υπάρχει επίση και δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό για την ανάπτυξη των επενδυτικών πολιτικών και των κατευθυντηρίων γραμμών, αλλά και την επιλογή των έργων. Και μια τελευταία παρατήρηση. Είμαι τη άποψη ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε η Επιτροπή Επενδύσεων να αποτελείται μόνο από οικονομολόγου. Η οικονομική πτυχή είναι μόνο μία από τι πτυχέ. θα προτιμούσα να έχουμε μια διεπιστημονική προσέγγιση, αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αναγκαίο, για την Επιτροπή Επενδύσεων και να βεβαιωθούμε ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια θα λαμβάνονται και αυτά υπόψη και θα ε, προωθούνται παρκού. Αυτή είναι μια επισκόπηση των σημαντικότερων παρατηρήσεων ε, σημείων τη γνωμοδότησή μα. Νομίζω ότι η πρόταση για το ΕΦΣΙ... Μας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουμε με τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, ώστε η οικονομία μας να ε, κάνει μια καλύτερη χρήση των πόρων. Εάν επικεντρωθούμε στις επενδύσεις που μπορούν να φέρουν τη διαφορά, μπορεί το ΕΦΣΥ να αλλάξει την οικονομία μας. Και να δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης. Αυτά από την πλευρά της ΕΝΒΗ. Είμαι σε επαφή και με τους εισηγητές της ε, ε, Επιτροπής Οικονομικών και της ΙΤΡΕ για να είμαστε βέβαιοι ότι η γνωμοδότηση της ΕΝΒΗ θα αντικατοπτρίζεται στο τελικό κείμενο για το ΕΦΣΥ. Πρέπει εν τέλει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη που κάνει σωστή χρήση των πόρων. Εάν όντω θέλουμε να ε, αναζωπηρωθεί η οικονομία μας και να δημιουργηθούν τέσσερις απασχόλησεις. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στους Κιώδης. Πρώτα απ' όλα από τα ΕΛΚ. Γκίζεκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Μίριαμ για αυτή την τόσο ισόρροπη προσέγγιση. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Η χρήση των δημοσιονομικών πόρων του Connecting Europe Facility και του Horizon 2020 ε, είναι κρίσιμη γιατί θα επηρεάσει την έρευνα και την κοινοτομία. Το Horizon 2020 λειτουργεί σωστά, είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξη για την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει βραχυπρόθεσμα με την ε, ε, λήψη κονδυλίων από αυτό να το αποδυναμώσουμε. Επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα έργα που θα επιλέγονται να προσελκύουν τους ιδιώτες επενδυτές, διότι θα πρέπει τα ποσά ε, που θα διατεθούν να ε, αντικατοπίζουν τους αρχικούς στόχους των... Ε, Επίσης να έχουν υψηλή κοινωνική αξία και να βοηθούν την βιώσιμη οικονομία. Πολλά, πολλές από τις τροπολογίες λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους στόχους, άρα θα τις υποστηρίξουμε. Όμως κάποιες τροπολογίες θα υποβάλω. Ιδιαίτερα για προγράμματα για καινοτόμες ε, υπηρεσίες υγείας. Εκεί υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Και επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε και προγράμματα δημόσιας υγείας γενικότερα. Γιατί η Ευρώπη θα μπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο μέλλον στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, e-health για παράδειγμα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ε, πιο φιλικές προς τις επενδύσεις ε, συνθήκες, ιδίως από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν απασχόληση. Άρα να μην ε, αυξήσουμε την γραφειοκρατία. Οπότε δεν υποστηρίζω την τροπολογία 8. Το ΕΦΣΙ δεν θα πρέπει να δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία. Θέλουμε αποτελεσματικότητα και όχι υπονόμευσή της. Οι δομές πρέπει να είναι όσο απλούστερες γίνονται, γίνεται. Και να μην έχουμε νέες εκθέσεις από πλευράς ε, εμπειρογνωμόνων κτλ. Το βασικό είναι οι εμπειρογνώμονες να μην είναι για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, αλλά για οικονομικά θέματα. Πρέπει λοιπόν το ΕΦΣΙ να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι η συγγήτρια όντως θα το βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Από τους συντεπτικούς που μεταρρυθμιστές, κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ σήμερα. Μιλώ εκ μέρους της κυρίας Γκίρλινγκ, η οποία είναι σκιώδης και σας ζητά συγγνώμη δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, εδώ, αλλά θα διαβάσω τις σημειώσεις της. Ο στόχο του ΕΦΣΙ είναι να υπάρξει μόχλευση για τι ιδιωτικέ επενδύσει, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να πετύχουμε μακροπρόθεσμα ανάπτυξη και ε, δημιουργία θέσεων εργασία. Η επιλογή των έργων λοιπόν θα πρέπει να είναι πάντοτε να χρησιμοποιήσει κριτήριο τη βιωσιμότητα των έργων βάσει επενδυτικών κριτηρίων. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα έργα αυτά έχουν μεγάλε πιθανότητε να πετύχουν του στόχου του Ταμείου, ε, μεταξύ των οποίων αυτοί που θα μεχλεύσουν τα μεγαλύτερα δυνατά ποσά ιδιωτικών επενδύσεων μεταξύ των υπόλοιπων που θα προταθούν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συγκεντρωθούν ε, τέτοιοι να συγκεντρωθεί για ποικιλία πιθανών έργων να επιλεγούν και μόνο βάσει τη πραγματική του αξία. Έχει βέβαια κάποιε δυσκολίε, κυρία Γκέλινγκ με το άρθρο 5 στι λεπτομέρειε των τροπολογιών, με την περιορισμό τη συγκέντρωση των έργων και τα πρόσθετα κριτήρια που προτείνονται. Εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο κατεξοχήν οικονομικό. Το να περιλάβουμε ε, υπερβολικά πολλά ε, περιβαλλοντικά κριτήρια θα μειώσει τον αριθμό επενδυτών που μπορεί να προτείνουν ε, έργα. Επιτέ, και μεταρρυθμιστέ έχουν κάποιε ανησυχίε για την πρόταση τη εισηγητρία να υπάρχει ένα περιβαλλοντικό εμπειρογνώμων και ένα κοινωνιολόγο στην Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επενδύσεων δεν πρέπει να λάβει πολιτικό χαρακτήρα ή να υπάρχει κάποια οποιαδήποτε προκατάληψη τομεακή. Η εντολή τη είναι πολύ σαφή. Οι συναλλαγέ να συμμορφώνονται με τι προδιαγραφέ που προβλέπει το άρθρο 5. Οπότε να μην υπάρχει ανα... δεν υπάρχει καμία ανάγκη να υποφέρουμε ότι η συμπερίληψη ενό περιβαλλοντολόγου ή ενό κοινωνιολόγου ε, θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτέ τι αρχέ. Επίση, η Γκίρλινγκ ε, βλέπει ότι δεν έχει καταφέρει να καλύψει το θέμα τη χρηματοδότηση η συγκεντρία. Η συγκεντρία στηρίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει 2,7 δι ευρώ από το Horizon 2020 και για να στηρίξουμε τι επενδύσει ε, γενικότερα στην οικονομία. Παρά το γεγονό ότι ένα μεγάλο μέρο του Horizon 2020 και των κονδυλίων του για την έρευνα, που κυρίω εξαρτώνται από την κρατική ε, βοήθεια, δεν θα είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΦΣΥ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να, έχουν, να υπάρχουν τεράστια περιβαλλοντικά ωφέλη από την περιβαλλοντική έρευνα στο μέλλον. Αλλά εάν ε, μειώσουμε τη συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα σήμερα, ε, μπορεί να διακυβεύσουμε τα μελλοντικά αποτελέσματα. Γι' αυτό οποιαδήποτε μείωση των κονδυλίων του Horizon 2020 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημαντική ε, συμβολή στην οικονομία τη πραγματική έρευνα, τη βασική έρευνα, προκαταρκτική που γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχουν βιώσιμα έργα που θα ε, επιζήσουν στην αγορά, ώστε ε, εφόσον να πάρουμε κονδύλια από το Horizon 2020, τουλάχιστον να υπάρξει μια αντιστάθμιση στην πραγματικότητα με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών. Ευχαριστούμε από του υπόλοιπου Σκιώδη. Δεν βλέπω εδώ τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι ο σκιώδης των Πρασίνων, οπότε θα συνεχίσω με την ε, συνεισφορά μου για την γνωμοδότηση περιέψη. να ευχαριστήσω και την συγγήτρια για το έργο της, την κυρία Ντάλη, αλλά και όλους τους συναδέρφους που πήραν το λόγο. Βλέπω ότι το σχέδιο έκθεσης, το σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον της κυρίας Ντάλη, αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στην κλιματική και ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μακροπρόθεσμους στόχους όπως είναι η ενεργειακή ε, απόδοση και πάρκια. Θέλω να τονίσω ότι όλες οι επενδύσει του Ευρωπαϊκού Αυτού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να καταλήξουν σε βιώσιμη οικονομία. Γι' αυτό και η Επιτροπή μας θέλει να πιέσει τις διαδικασίες ώστε το Ταμείο αυτό να μην στηρίξει έργα τα οποία να κάνουν ζημιά στο περιβάλλον. Τώρα για τα προτινόμενα έργα. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα πρέπει να λαμβάνονται με απόλυτη διαφάνεια και αυτοί που τις παίρνουν να λογοδοτούν. Μερικές φορές έχουμε πρόβλημα από αυτού. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, τον εφοδιασμό δηλαδή, οι άλλες περιπτώσεις δεν βλέπουμε να υπάρχει διαφάνεια στις αποφάσεις. Δεν καταλαβαίνουμε πώς αποφασίζεται και πώς επιλέγεται το κάθε έργο. Γι' αυτό στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Αυτού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων θέλουμε πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής. Τώρα, η εκτίμηση κινδύνου. Όλοι ξέρουμε ότι θα υπάρξουν εγγυήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Όμως πρέπει να αποφύγουμε κίνδυνος ιδιωτικών επενδύσεων να περνάνε στους ώμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Πρέπει να πρόκειται για βιώσιμα έργα που θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή των έργων που να είναι βιωσιμότητα. Αν δεν μπορούμε να υπάρχουν άλλα κριτήρια, να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Συγκεκριμένα κριτήρια λοιπόν είναι κάτι αναγκαίο. Όσον αφορά για τη στρατηγική επενδύσεων στο μέλλον, τα εφή δίκτυα, αποθήκευση, νομίζω ότι όλες οι επενδύσεις για την ενέργεια πρέπει να βάζουν πρώτα απ' όλα την εξοικονόμηση. Την επάρκεια και την αύξηση του ποσοστού εναλλακτικών πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Τα έργα επίσης πρέπει να ελέγχονται ανάλογα με τα αποτελέσματά τους στην βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Πολύ συχνά είναι κάτι που δεν το βάζουμε στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική διοπικιλότητας δεν πετυχαίνει πάντα τους στόχους της. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και αυτό ως κριτήριο. Τέλος, προτείνω στον κατάλογο του άρθρου 5 να βάλουμε και την βιώσιμη διαχείριση. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο Βιώσιμη διαχείριση υδάτων λοιπόν. Πρέπει και αυτό να συμπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό στο 5. Και εγώ λοιπόν προσβλέπω σε καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και με τους υπόλοιπους όδες εισηγητές. Και τώρα περνάμε στο EFDD. Η Ελεονόρα έδειχε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συνάδελφο Νταλή για την πρότασή της. Μια προκατακτική παρατήρηση. Λείπουν οι επενδύσεις. Το λέει και ποτάς κανονισμού. Η προοπτική αυτή οφείλεται και στι διορθώσεις περί προπολογισμού και τις πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν τα κρατημέλη τα τελευταία χρόνια. Αυτά συνέχληψαν τη ζήτηση και έχουν διωγγώσει την αβεβαιότητα. Είναι λοιπόν σαφές ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι πολιτικές λιτότητες για να υπάρξουν επενδύσεις. Από το πρόγραμμα επενδύσεων, όπως το προτείνει η Επιτροπή, θα μπορούσε να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για όλες τις δραστηριότητε. που ίσως να στήριζαν οι επενδυτές παρά τον κίνδυνο. Όμως, τον κανονισμό δεν προβλέπονται μέσα για την αποσύνδεση μεταξύ ε, οικονομικής ανάκαμψης και περιβαλλοντικού αντικτύπου, δηλαδή χρήση των πόρων. Επί χρόνια η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο ε, μας ζητά να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση στηρίζοντας την πράσινη και την κυκλική οικονομία. Τώρα έφτασε η στιγμή να δράσουμε επιτέλους. Και όχι μόνον οι δραστηριότητες της πράσινης οικονομίας είναι πιο ε, επικίνδυνες από οικονομικής πλευράς, αλλά είναι και αυτές που θα πρέπει να περάσουν ακριβώς στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου. Επίσης, η διάσταση της καινοτομίας και από την ε, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μεταξύ των μεγάλων υποδομών που χρειάζονται για τη στήριξη της ανάπτυξης, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί την παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο για την ε, πρόληψη φυσικών καταστροφών, την ξηρασία, την λειψιδρία, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές. Η μεγάλη δηλαδή υποδομή που πρέπει να ε, προάγουμε είναι αυτό που αφορά την προστασία της επικρατειάς μας, των ε, επιμέρους περιοχών. Δεν είναι απλώς οι υποδομές και οι επενδύσεις που έχουν να κάνουν και πάλι με τη χρήση με την χρήση, την αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μόνον. Ως προς τα την Επιτροπή Επενδύσεων θεωρούμε ότι είναι περιττή η δημιουργία τους. Τη λειτουργία αυτή μπορούν να την αναλάβουν οι υπεύθυνοι της ΕΤΕ χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν και άλλα ποσά για τη δημιουργία νέας δομής, νέας ομάδας. Και πρέπει να βουλευτούν και διαδικασίε, ώστε όλη η διαδικασία επιλογή των έργων, αλλά και η έγκρισή του και η εξολογή των αποτελεσμάτων να είναι διαφανή, διαφανής και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και συμμετοχή των πολιτών είτε των ομονωμένων πολιτών είτε οργανωμένων σε ενώσει συλλογικού συμφέροντο. Μια τελευταία αναφορά. Οι εταιρείε, οι οποίε αναφέρονται στο κείμενο, οι οποίε θα αποφυληθούν από τη χρηματοδότηση, ε, αναφέρονται ως 300, ε, αυτές που έχουν ως 300 ε, μισθωτούς. Ε, μα εδώ μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ελάχιστες επιχειρήσεις και αυτές που είναι νεοφυείς και καινοτόμες. Αυτές θα πρέπει να στηρίζουμε. Να, καταλα... να μειώσουμε λοιπόν τον ε, αριθμό των 3.000 υπαλλήλων. Νομίζω ότι ξεφεύγουμε από τις πραγματικές απαιτήσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες κάνονται να καλύψουμε. Και που κατά τα άλλα από τον ίδιο τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν τους 250 υπαλλήλους. Τεράστια διαφορά. Ευχαριστώ. Thank you and... Ευχαριστώ. Και από ό,τι έμαθα, ε, ο κύριος Πέτερ αντικαθιστά το σκιώδη, ή η κυρία Πέτερ, αντικαθιστά το σκιώδη της Άλντε. Ζητά συγγνώμη ο σκιώδης μας, ε, στηρίζουμε την εισηγήτρια και να προσθέσω τα εξής. Είμαστε υπέρ εναλλακτικής χρηματοδότησης Για παράδειγμα, ποσά που δεν έχουν αξιοποιηθεί στο τέλος του χρόνου από διάφορα ταμεία. Αυτά θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε, να αλλάξουμε το σύστημα. Και αν το κάναμε αυτό δεν θα χρειαζόταν να αφαιρέσουμε πόρους από τον ορίζοντα 2020 και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη ιδιαίτερα τον ορίζοντα 2020 που κάναμε τόση προσπάθεια κατά την προηγούμενη θητεία για να του δώσουμε αρκετή πρικοδότηση και θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε τεχνολογίες εχμής ούτως ώστε να διατηρήσουμε την πρωτοπορία μας από πλευράς επιστημονικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων. Βεβαίως ε, καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους ε, δημιουργείται αυτό το νέο ταμείο από πλευράς του Γιούνκερ. Αλλά εκτός αν ε, είναι επιθεία και ξέρει τι ακριβώς θα επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα, πώς μπορεί να θεωρήσει ότι αφαιρώντας πόρους από το ορίζοντα 2020 δεν θα θίξει τους στόχους μας αντί να τους προωθήσει. πρέπει ό,τι επιχειρούμε να είναι βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Και επίσης πρέπει να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες με απλές και αποτελεσματικές και ταχύ διαδικασίες. Δεν πρέπει να χρηματοδοτούμε αυτά τα προγράμματα που δεν αποδίδουν και κρατάνε πολλά χρόνια. Ξέρετε τι εννοώ. Και πρέπει να υπάρχουν και επαρκείς μηχανισμοί για να ε, υπάρχει η αναγκαία λογοδοσία. Είναι δημόσιοι οι πόροι, πρέπει λοιπόν να δαπανώνται με διαφανή τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπέζα. Και τώρα συνάδελφοι. Πρώτος ο κύριος Μπάλας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να χαιρετήσω τη δουλειά της εισηγητρίας της κυρίας Νταλή. Και κυρίως να σταθώ στην ε, παρατήρηση του σκιώδησου και του, των συντηρικών και μεταρρυθμιστών αλλά και των σοσιαλιστών και δημοκρατών για την ε, αφιβολία που έχουμε σήμερα για την ε, σύνθεση Τη σύνδεση τη Επιτροπή Επενδύσεων, όπω την προτείνουμε εμεί σήμερα, για να υπάρχουν και άλλοι εμπειρογνώμονε. Γιατί να βάλουμε κοινωνιολόγο ή περιβαλλοντολόγο στην Επιτροπή αυτή, για να έχουν μια φωτισμένη τοποθέτηση για την επιλογή των προγραμμάτων και με την χρηματοδότηση, την επιλογή των έργων και τη χρηματοδότησή του και για να την υπάρχει περισσότερο γραφειοκρατικό άρθρο. Δεν είναι αυτή ο που δημιουργεί γραφειοκρατικό άρθρο σε αυτή την περίπτωση. Δεν θέλω να στιγματίσω κανέναν βέβαια, τους περιβαλλοντολόγους, τους κοινωνιολόγους λέγοντας ότι είναι πιο γραφειοκράτες από άλλους όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε παρόμοια ε, συμπεριφορά ω προς τις επενδύσεις και βλέπουμε ότι όταν υπάρχει οικονομική μονοδιάσταση στι επενδύσεις πολλέ φορές ο στόχος δεν επιτυχάνεται. Δεν λαμβάνει υπόψη τα λεπτά χαρακτηριστικά των ε, αναγκών των τοπικών ή τις γνώσεις, τις δεξιότητες των εργαζομένων ή την, το εύστοχο, το περιβαλλοντικό και το τοπικό ε, ε έργου, μιας επιλογής. Γι' αυτό λοιπόν καλό να σκεφτούμε για το θέμα αυτό πολύ προσεκτικά για να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί οι επενδύσεις δεν είναι απλώς ε, χρηματοπιστωτικό ή οικονομικό ζήτημα πλέον σήμερα. Κατά τα άλλα συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να προσπιστούμε σήμερα το Horizon 2020 ως ένα από τα προγράμματα που και σταθερό είναι και που δεν νομίζω ότι η κυρία Ανταλή σήμερα θέλει να προτείνει να πάρουμε από εκεί κοντήλια για να στηρίξουμε το ΕΨΙ. Δεν το είπε καν άλλωστε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε έναν αγώνα κοινό για όλο το κοινοβούλιο που και θα διεξαχθεί και αν ε, βρούμε εναλλακτικές λύσεις τόσο το καλύτερο. Και μια ακόμη παρατήρηση για τις τροπολογίες που θα υποβάλω, κυρίως για τις ιδεολογικές σκέψεις που αφορούν το όλο πρόγραμμα, όχι το σχέδιο γνωμοδότησης, δεν είναι αυτό, ενώ το ΕΦΣΥ, θα πρέπει να προσέξουμε να μην συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπληκτική μακροοικονομική πολιτική που έχει σχεδιάσει και ακολουθήσει στο παρελθόν. Θα πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και ειλικρινείς ως προς τις αποτυχίες του παρελθόντος. Uh, Ευχαριστούμε. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξέρετε ότι πολύ χαίρομαι όταν μιλάμε για την Ολλανδία και πολύ θέλω να ξέρω τι θα γίνει με τα έργα τα σχετικά. Χαίρομαι λοιπόν που άκουσα τέτοια πράγματα και θέλω να ξέρω πώς θα νιώσει ο κάθε Ευρωπαίος ότι γίνονται έργα για αυτόν και όχι για τις πολυεθνικές. Αυτό είναι το σήμα που πρέπει να στείλουμε για την ψηφιακή ατζέντα τώρα. Πρόκειται για την υγεία, πρόκειται για τους ηλικιωμένους στην Ήπεθρο, σε συνδυασμό με τους γιατρούς, για την Ήπεθρο, πρόκειται για τους αγρότες, οι οποίοι θέλουν κάποια βοήθεια, θέλουν συνεργασία. Θέλω να πω ότι υπάρχει τεράστιος δυναμισμός και Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία να αρχίσουμε. Δεύτερον, για άλλα προγράμματα, μεγάλα προγράμματα του Ταμείου αυτού, του Ευρωπαϊκού Ταμείου, πρέπει να δούμε και το θέμα των ουδέτερων λεγόμενων κατοικιών ενεργειακά. Πώς χτίζονται, πώς μπορεί να χτίσει ένας οικοδόμος τέτοια σπίτια. Τέτοια έργα πιστεύουμε ότι είναι επίσης πολύ θετικά. Και θέλω να δω πώς θα προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Μπάρτσο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η εισηγήτρια έχουμε τώρα τις τροπολογίες από την εισηγήτρια Νομίζω ότι έχει υπερβολικές ε, προσδοκίες από αυτό το ταμείο. Εγώ είμαι λιγάκι πιο επιφυλακτικός για αυτό το θέμα. Έχω θέσει τα ζητήματα που με ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα το ποσό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει με 21 δις και λέει ότι θα έχουμε έναν πολλαπλασιαστή 15. Μα τι είναι αυτό, είναι θαύμα αυτό. βιβλικό σχεδόν, σχεδόν. Χρειάζεται να έρθει ο Ιησούς για να ταΐσει τόσο πολλούς. Πώς θα πείσουμε τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει. Βεβαίως, είναι πολύ ελκυστικό για τους ε, ιδιώτες επενδυτές να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις από το δημόσιο κορβανά. Αλλά στην Ουγγαρία έχουμε πολύ αρνητική εμπειρία με τα λεγόμενα PPP, δηλαδή τις ε, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και αν κατάλαβα καλά, ε, και ο εισηγητής, ο σκιώδης των Πρασίνων είπε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο. Ένας μεγάλος κίνδυνος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τελικά να πληρώσει πάλι τα σπασμένα ο φορολογούμενος. Και κάτι ακόμη. Η συγκήτρια μας είπε ότι ο πρώτος στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ένωση γύρω στο 75% ε, είναι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι πρέπει να προωθήσουμε κυρίως τις μικρομεσαίες. Αλλά τι λέει το κείμενο. Η Τράπεζα Επενδύσεων, εκεί που λέγεται ότι η Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να τα στηρίξει όλα αυτά, ότι οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν ε, στο προσκήνιο τις μικρομεσαίες και μετά στην επόμενη παράγραφο λέει ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως, κατά πρώτο λόγο, έως 3.000 εργαζομένους. Μα τι μικρομεσαίες είναι αυτές. Ο κανονικός μας ορισμός λέει ότι είναι μικρομεσαίες αν έχουν μέχρι 250. Αυτό είναι μια σαφής αντίφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκπρόσωπος της Επιτροπής. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πει τίποτα. Η κυρία Μαλίνα Μάζαν από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ. Παρακαλώ. Πείτε μας την άποψή σας για την γνωμοδότηση και τις απόψεις των σκιωδών. Η κυρία Μάτσον. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμμετοχή της Επιτροπής σα στο και σας ευχαριστώ για την ταχύτητα με την οποία ε, αντιμετωπίζετε αυτό το σημαντικό θέμα συναπόφασης. Το γεγονό το θεωρείτε ως πολύ σημαντικό νομίζω καταδεικνύεται και από την ενασχόληση τόσο πολλών επιτροπών. Αυτό θέτει κάποια προβλήματα για το χρονοδιάγραμμα. Αλλά η Επιτροπή χαίρεται που τόσο πολλές επιτροπές ε, ασχολούνται και λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας λέτε. Για το θέμα του προπολογισμού, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάργηση των άρθρων 18 και 19 που προτείνουν κάποιες επιτροπές. Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για τον προπολογισμό της Ένωσης και γι' αυτό έχουμε υποβάλει αυτή την πρόταση. Να μην καταλήξουμε να συζητάμε κάθε χρόνο το θέμα αυτό, και πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου για να προσελκύσουμε τους ιδιώτες επενδυτές και να έχουμε αυτό το μοχλευτικό αποτέλεσμα στο οποίο βασίζεται το ΕΦΣΙ. Πρέπει να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση. Η συμβολή από τον ορίζοντα και το Συνδέοντα στην Ευρώπη δεν είναι χαμένα λεφτά. Έτσι θα έχουμε σημαντικές επενδύσεις που θα επενδυθούν στην καινοτομία. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τις χρηματοδοτήσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε τις επενδύσεις και στις υποδομές και στην καινοτομία. Πιστεύω ότι μέσω αυτής της ε, διαφορετικής χρήσης των χρηματοδοτήσεων του ορίζοντα και του συνέδρα στην Ευρώπη θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η προσθετικότητα επίση αναφέρθηκε από ορισμένου. Βεβαίω, ακρογωνία λήθο τη πρότασή μα. Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτούνταν από τον ιδιωτικό τομέα ή το δημόσιο με λογικού όρου, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ. Η ανεξαρτησία τη Επιτροπής Επενδύσεων για να αποτιμήσει την προστατικότητα και οι τακτικές ε, υποβολές εκθέσεων θα διασφαλίσουν ότι τα κριτήρια αυτά θα γίνουν σεβαστά. Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι ακρογωνία λίθος της πρότασης, το είπα και προηγουμένω. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη χρηματοδότηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πρέπει να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικού επενδυτέ για να επιτύχει το ΕΦΣΥ. Άρα πρέπει να είναι εντελώ αποπολιτικοποιημένο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να εμπλακεί άμεσα με την Επιτροπή Επενδύσεων, ούτε η Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή επενδύσεων θα αποτελείται από ανεξάρτητους ειδήμονες που θα εφαρμόζουν τις καθευντήρες γραμμές που βέβαια έχουν ε, αποφασιστεί και με πολιτικά κριτήρια. Είχατε σχόλια και για αυτές λοιπόν τις καθευντήριες. Βασικό είναι να είναι εύχριστες και ευέλικτες αυτές οι καθεντήρες. Αλλιώς θα πνίξουν τις προσπάθειες. Η Επιτροπή δεν στηρίζει τομεακές ή γεωγραφικές χρηματοδοτήσεις, δηλαδή κατανομές χρηματοδοτήσεων. Αυτή η ευελιξία πρέπει να διατηρηθεί. Θα υποβάλουμε τακτικά εκθέσεις ετησίως, ε, ενδιάμεσες εκθέσεις. Άρα θα συνεχίζετε να έχετε δυνατότητα να ελέγχετε ότι τηρούνται τα κριτήρια που θα έχουν καθοριστεί για τις μελέτες αντικτύπου. Ορισμένα από τα προγράμματα από τα οποία θα εστιάσει το ΕΦΣΥ θα είναι πολύ μικρά βεβαίως. Άρα να το λάβουμε υπόψη όταν ε, επιβάλλουμε τέτοιες υποχρεώσεις σε τόσο μικρά προγράμματα. Μπορεί να είναι υπερβολικό. Τέλος, παρακολουθούμε στενά τις εργασίες επ' αυτού και όλων των άλλων επιτροπών και προσβλέπουμε, προσβλέπουμε στην τελική σας γνωμοδότηση και την ε, τελική έκθεση του Κοινοβουλίου για να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ντάλη, η συγκήτρια. Ευχαριστώ τους ε, σκιώδεις, όλους τους συναδέλφους. Φαίνεται ότι συνολικά συμφωνούμε για τα βασικά θέματα που έχουν ε, μεγάλη σημασία για την ΕΜΒΗ. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που θέλω να διευκρινίσω. Το θέμα των κατοφλίων, δηλαδή ανώτατος αριθμός εργαζομένων. Θέλουμε χαμηλότερο επίπεδο. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα που το συζητάει και η ΕΚΟΝ. Στην έκθεσή της. Κάτι άλλο για τα θετικά κριτήρια. Ερώτημα. Αν η ΕΝΒΗ δεν πιέζει για να υπάρχουν βιώσιμα προγράμματα και ενεργειακά αποδοτικά, ποιος θα το κάνει. Η δική μας Επιτροπή προωθεί αυτά τα θέματα και είμαι πεπισμένη ότι το περιβάλλον <clears throat> και η οικονομία μπορούν να συμβαδίσουν. Και δεν νομίζω ότι να απαιτήσουμε φιλικά προς το περιβάλλον προγράμματα σημαίνει ότι διώχνουμε τους επενδυτές. Δεν το πιστεύω. Αντίθετα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε πιο πράσινη οικονομία. Το περιβάλλον και η οικονομία μπορούν να συμβαδίσουν. Άλλο που ετέθη έγινε μια δήλωση ότι φαίνεται ότι η συγγήτρια είναι υπέρ του να φερθούν 2,7 από το συνδέοντα στην Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020. Αβάσιμος αυτός ο ισχυρισμός. Και να διευκρινίσω ότι εννοώ. Η χρηματοδότηση από τον ορίζοντα και το συνδέοντα στην Ευρώπη Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας της Ήτρε. Και η Ήτρε λέει ότι η συμβολή του ενωσιακού προπολογισμού θα πρέπει να εγκριθεί σταδιακά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα πλαίσια τη ε, διαδικασία έγκριση του προπολογισμού έω το 2020. Και η αρχή του προπολογισμού θα χρησιμοποιήσει όλου του ε, ισχύοντε μηχανισμού ευελιξία αντί να πάρει από τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα. Θέλω λοιπόν να σα διαβεβαιώσω ότι σε τελευταία ανάλυση αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω αυτή τη γνωμοδότηση είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργήσει σωστά το ΕΦΣΙ. Και τέλος, τέλος, για την Επιτροπή Επενδύσεων. Πρέπει να είναι πιο ποικιλόμορφη. Να μην έχει μόνο ε, εμπειρογνώμονες για χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν τα επιτύχαμε τόσο καλά. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτή την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουν όλοι ε, γνώσει στον ίδιο τομέα σε αυτήν την Επιτροπή. Πρέπει να έχουν γνώσει σε διαφορετικού τομεί. Γιατί αλλιώ η όλη προσπάθεια δεν θα αποδώσει. Σα ευχαριστώ όλου του κοιόδη και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μαζί σα γιατί ο στόχος μου είναι η γνωμοδότησή μας να είναι αποφασιστική και να προωθήσει τις απόψεις μας για το ΕΦΣΙ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο σημαντική σας δήλωση. Να περάσουμε στο χρονοδιάγραμμα του όλου θέματος. Είναι αρκετά πιεστικό. Θεσμό για την υποβολή τροπολογιών 23 Μαρτίου 6 το απόγευμα επόμενη εβδομάδα ψηφοφορία στην ΕΝΒ στις 14 Απριλίου Πρώτο σημείο, ίσως και όλα στην ημερήσια διάταξη, κατά τις 9 το πρωί. Ε, ψηφοφορία στις Επιτροπές οίκων και Budget στις 20 Απριλίου. Και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Και πάλι ως τελευταίο σημείο να θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και 30-31 Μαρτίου και πάλι στις Βρυξέλλες. Και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.